Um, Συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε παρακαλώ. Είναι εδώ ο κύριος Μπόνι για το πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης, η οποία είναι πολύ βεβαρημένη. Στις 10.45 θα έχουμε την παρουσίαση της Λετωνικής Προεδρίας και θέλω να είμαι δίκαιος έναντι των συναδέλφων που ήρθαν εδώ στις 9 και δεν έχουν καθυστερήσει. Ζητώ συγγνώμη λοιπόν για την καθυστέρηση των 7 λεπτών. Ξεκινάει η συνεδρίασή μας. Καθυστερήσαμε λίγο να ξεκινήσαμε, να ξεκινήσουμε γιατί θέλαμε να δούμε αν, αν λειτουργεί το PowerPoint και δυστυχώς δεν λειτουργεί. Εν πάση περιπτώσει ας προχωρήσουμε αν συμφωνείτε. Πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης για τα ναρκωτικά και την τοξικομανία. Θα έχουμε παρουσίαση από τον Διευθυντή, κύριο Wolfgang Goetz, παρουσίαση της έκθεσης για τα ναρκωτικά στην Ευρώπη το 2015, τάσεις και εξελίξεις. Σας καλωσορίζω κύριε Goetz, χαίρομαι πολύ που είστε εδώ στις Βρυξέλλες για να μας παρουσιάσετε την έκθεσή σας. Να σας δώσω το λόγο για 10 λεπτά περίπου και μετά θα ξεκινήσει η συζήτηση. Ζητώ συγγνώμη όμως που το PowerPoint δεν είναι διαθέσιμο. Ε, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Yeah, thank you, uh, and Ευχαριστώ κύριε ε, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί σας. Είναι η ενδέκατη φορά που ε, παρουσιάζω την ε, έκθεση για τα ναρκωτικά στην Ευρώπη. Έχω έρθει πολύ περισσότερες φορές εδώ και χαίρομαι διότι μπορώ να σας ε, παρουσιάσω την ανάλυση που κάνουμε για την κατάσταση στην Ευρώπη. Επιτρέψτε μου δύο γενικές παρατηρήσεις να κάνω καταρχάς. Πρώτον, την Παρασκευή με μήνυμα ηλεκτρονικό ταχυδρομείου σας στείλαμε την ε, έκθεση για το 2014 και θα δείτε τα επιτεύγματά μας για την προηγούμενη χρονιά. Εάν έχετε ερωτήσεις για το email που λάβατε και την έκθεση, ευχαριστώ να απαντήσω σήμερα σε άλλη συνεδρίαση ή με mail επίσης. Αυτό καταρχάς. Κατά δεύτερο, να σας ευχαριστήσω για τη στήριξή σας, γιατί καταφέραμε ε, τον προϋπολογισμό του Κέντρου Παρακολούθησης του Παρατηρητηρίου να τον προσαρμόσουμε στο αυξημένο φόρτο εργασίας μας. Εσείς ψηφίσατε τροπολογίες για την αύξηση του προϋπολογισμού, τις οποίες ε, επικύρωσε η Επιτροπή ε, για τον έλεγχο του προπολογισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις οποίες ενέκρινε όλο το Κοινοβούλιο, δυστυχώς όμως χάθηκαν με τη συνδιαλλαγή από πλευράς ε, Συμβουλίου. Εάν όμως με στηρίξετε φέτος, ε, θα προσπαθήσουμε ξανά. Ολοκληρώνεται η εντολή μου στα τέλη αυτής της χρονιάς, αλλά εάν τα καταφέρουμε δεν θα επανέλθω με αυτό το ζήτημα να σας το ζητώ ξανά και ξανά. Ας επανέλθουμε τώρα στην κατάσταση των ε, θεμάτων που μας απασχολούν. Είναι η 20η ανάλυση που κάνουμε για το πρόβλημα με τα ναρκωτικά στην Ευρώπη και ε, το, οι δέσμοι εκθέσεων που σας στείλαμε σήμερα ε, δεν έχει πολλές ομοιότητες με την πρώτη έκθεσή μας του 1996. Το 1995 όταν ξεκινήσαμε να, να δουλεύουμε με 15 κράτη-μέλη ήταν επιδημία ηρωίνης τότε εκείνη την εποχή. Το βασικό πρόβλημα ήταν η μετάδοση του AIDS και η χρήση ηρωίνης. Οι απαντήσεις που χρειάζονται σε αυτό το πρόβλημα υπάρχουν ήδη, αλλά έχουν προκύψει άλλα ζητήματα που απαιτούν την προσοχή μας. Η ηρωίνη είναι υπεύθυνη για μεγάλο μέρος των προβλημάτων που σχετίζονται με τα ναρκωτικά στην Ευρώπη. Ωστόσο, οι τελευταίες εξελίξεις στο θέμα αυτό είναι θετικές. Η μείωση των χρηστών ηρωίνης είναι εμφανής. Από το 7 μέχρι σήμερα οι ηρωνομανείς που ζητούν θεραπεία και απεξάρτηση έχουν μειωθεί στο μισό, ενώ όλοι οι δείκτες σε σχέση με τη ηρωίνη έχουν μειωθεί. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην Ευρώπη είναι ότι το 1,3 εκατομμύρια χρήστες αυτή τη στιγμή έχουν ε, σήμερα είναι σε προγράμματα υποκατάστασης. Η ηρωινοεξάρτηση είναι μια χρόνια κατάσταση και θα πρέπει οι υπηρεσίες να προσαρμοστούν στις ανάγκες των χρηστών οι οποίοι γυράσκουν. Και όλα αυτά περιπλέκονται από το ότι γίνεται κακή χρήση των βενζοδιαζεπινών και έτσι υπάρχει αυξημένος ε, κίνδυνος ε, ε, overdose, θανάτου από υπερβολική δόση. Είχαμε πάνω από 2.000 θανάτους τέτοιου είδους στην Ευρώπη το 2013 και τώρα έχουμε ε, ε, εκπαίδευση, προγράμματα εκπαίδευσης και των χρηστών και των ιατρών για τα συμπτώματα και τις καταστάσεις που έχουν να κάνουν με την υπερβολική ε, δόση, με το overdose. 1.500 διαγνώσεις ε, ε, φορέων του AIDS στη Ρουμανία ετησίως είναι το μικρότερο ποσοστό σε μία δεκαετία. Όμως έχουμε υψηλά ποσοστά υπατήτηδας σε, σε αυτό τον πληθυσμό. Και τώρα διατίθενται αντιοικά ε, φάρμακα όλο και περισσότερο στους φορείς υπατήτηδας σε. Ωστόσο το κόστος είναι πολύ ψηλό και αυτό, είναι, ε, αυτό προκαλεί ανησυχία. από το 2009 ο αριθμός των χρηστών ηρωίνης έχει μειωθεί. Οι 5,6 τόνοι ηρωίνης που έχουν κατασχεθεί το 2013 είναι από τα χαμηλότερα και τα λιγότερα φορτία των τελευταίων 10 ετών, ωστόσο οι ανησυχίες παραμένουν. Πρώτον, έχει αυξηθεί σημαντικά η οπιοπαραγωγή στο Αφγανιστάν. Είναι η χώρα που προμηθεύει την ηρωίνη στην Ευρώπη σε μεγαλύτερο βαθμό και έχει και δυνατότητες να προσφέρει και να έχει διαθεσιμότητα ηρωίνης και στο μέλλον. Από εκεί και πέρα έχουμε ανοιχνεύσει δύο εργαστήρια επεξεργασίας της ηρωνίας στην Ισπανία και υπάρχουν και αλλαγές στους δρόμους, στις διαδρομές με τις οποίων έρχονται τα ναρκωτικά ηρωίνη στην Ευρώπη. Τα προβλήματα που σχετίζονται με τη χρήση της κάναβης αυξάνονται. 60.000 άνθρωποι για πρώτη φορά αναζήτησαν θεραπεία απεξάρτησης από την κάναβη το 2013, ενώ είναι το πιο διαδεδομένο παράνομο ναρκωτικό στην Ευρώπη. 20 εκατομμύρια ενήλικες χρησιμοποίησαν κάναβη την περασμένη χρονιά, ενώ το 1% όλων των ενηλίκων Ευρωπαίων χρησιμοποιεί κάναβη καθημερινά. Γίνονται και υπάρχουν πρωτοβουλίες για να ρυθμιστεί η πώληση της κάναβης στη ΣΥΠΑ και αλλού, ενώ στην Ευρώπη εστιαζόμαστε κυρίως στο θέμα του κόστους. Και γι' αυτό θεωρούμε ότι παραμένει η αρμοδιότητα των αρχών επιβολής του νόμου. για το ε, ε, είναι το 63% των, αδικη... των αδικημάτων που διαπράττονται ε, σε σχέση με τα ναρκωτικά στην Ευρώπη, τα οποία είναι συνολικά 1,2 εκατομμύρια. Έρχομαι τώρα στην κοκαίνη και στην μεταμφεταμίνη. Είναι η κοκαίνη το πιο ευρύ διεγερτικό στην Ευρώπη. 2,5 εκατομμύρια ενήλικες το χρησιμοποιούν. 1,8 εκατομμύρια χρησιμοποίησαν έκσταση και 1,3 περίπου αμφεταμίνες. Η χρήση όλων αυτών σταθεροποιείται ή μειώνεται. Η ένεση μεθαμφεταμίνες και άλλων από, ε, ε, δημιουργούν προβλήματα σε συγκεκριμένες ομάδες χρηστών, σε συγκεκριμένες χώρες. Βεβαίως είναι προφανή τα προβλήματα με τη χρήση κοκαίνης, χασής, ηρωίνης κτλ. σε σχέση με την περιεκτικότητά τους και την όθευσή τους έχουν αυξήσει το μερίδιο της αγοράς τους άλλα προϊόντα φυτικά που υποκαθιστούν την κάναβη. Έχουμε το χασίς, το οποίο μάλλον συνδέεται με νέες πρακτικές του Μαρόκο. Από πλευράς καθαρότητας, Τώρα έχουμε περισσότερα δισκία ε, έκσταση και με την Europol έχουμε προειδοποιήσει δημόσια για τους κινδύνους κατανάλωσης τέτοιων προϊόντων. Μετά από σειρά θανάτων ε, υπήρξε δημόσια προειδοποίηση για δισκία και ταμπλέτες ε, έκσταση που είχαν και άλλες βλαβερές ουσίες όπως το PMMA. Η τεχνολογική καινοτομία και ο ανταγωνισμό τη αγορά είναι τα δύο στοιχεία που ευθύνονται για την όλο και μεγαλύτερη και περισσότερη καθαρότητα των ναρκωτικών που μπαίνουν στην αγορά. Για πρώτη φορά έχουμε δεδομένα και κατασχέσεις των φορτίων, άρα ε, προγραμματίζονται οι εισαγωγές τέτοιου είδους ουσιών για να αποτελέσουν μέρος των συνθετικών ναρκωτικών. Η διαθεσιμότητα όλων αυτών ε, παίζει σημαντικό ρόλο. Σε κάποιες αγορές πραγματική εναλλακτική στη κάναβη ε, ή στα ναρκωτικά χαμηλής ποιότητας είναι η συνθετική κάναβη και συνθετικά ναρκωτικά που είναι στο εργαστήριο ε, που έχουν καφεϊνοειδείς ουσίες. Τώρα παρακολουθούμε πάνω από 400 νέες ουσίες, τέσσερις φορές περισσότερες από ό,τι πριν από τέσσερα χρόνια. Έχουμε 101 νέες ουσίες που ανοιχνεύσαμε πέρσι, 31 καφεϊνοειδή και άλλα τόσα περίπου καναβιδο, καναβινοειδή. Όλα αυτά είναι, υποκαθιστούν τα διεγερτικά ε, και τα συνθετικά ναρκωτικά και, την, και το έκσταση. 61% των 35.000 κατασχέσεων ψυχοδραστικών ουσιών του 2013 ήταν το 61% καφεϊνοειδή. Στις περισσότερες νέες χώρες η επικράτηση αυτών των νέων ουσιών είναι χαμηλή, όμως έχουν πάρα πολύ ψηλή τοξικότητα, ορισμένες ψυχοδραστικές ουσίες, και ακόμα και η περιορισμένη χρήση δημιουργεί ανησυχίε και προβλήματα. Η πολύ περιορισμένη χρήση. Κυρίε και κύριοι, η νέα Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Ασφάλεια αναγνωρίζει το πρόβλημα των ναρκωτικών, τι συνδέσει του με το οργανωμένο έγκλημα, με το, την καινοτόμο αγορά πραγματικά στην παραγωγή και πώληση των ναρκωτικών. Το σύστημα παρακολούθησης που έχουμε λοιπόν εμείς πρέπει να εξελιχθεί για να μπορεί να παρακολουθεί τις αλλαγές και να δίνει έγκυρα στοιχεία για να ληφθούν σωστές αποφάσεις. Τα τελευταία 20 χρόνια η πολιτική για τα ναρκωτικά απομακρύνεται από την ιδεολογία και προσεγγίζει όλο και περισσότερο τα στοιχεία. Και γι' αυτό είχαμε επιτυχία ε, για, ε, όταν εισαγάγαμε τις, ε, τα δημοκρατικά δικαιώματα τις έννοιες της ελευθερίας και της δημοκρατίας στην καταπολέμηση των ναρκωτικών. Η το ΟΥΝΚΑΣ 2016 πλησιάζει. Είναι η συνεδρίαση των Ηνωμένων Εθνών για το πρόβλημα των ναρκωτικών παγκοσμίω και πρέπει όλοι να μιλήσουμε εκεί με μία φωνή για να ε, υπάρξει περισσότερη ευρωπαϊκή χρειά στην πολιτική καταπολέμηση των ναρκωτικών και στι άλλε περιοχέ του κόσμου. Θα πρέπει να συμβάλλουμε στι πολιτικέ αποφάσει και να ενημερώσουμε το κοινό και στι άλλε χώρε και εκτό Ευρώπη, όπω κάνουμε εμεί εδώ τα τελευταία 20 χρόνια. Είμαι βαθιά πεπισμένο ότι για να είναι πιο αποτελεσματική η πολιτική των ναρκωτικών μας στο μέλλον πρέπει να βασιζόμαστε περισσότερο στα στοιχεία και η Ευρώπη πρέπει να είναι πολύ πιο παρούσα και ισχυρή διεθνώς. Ευχαριστώ πολύ. Um, so our joint rapporteurs the ongoing proposal. Ευχαριστώ, ευχαριστούμε για την παρουσίαση αυτή. Θα καλέσω και τους δύο συνεισηγητές να πάρουν το λόγο για το θέμα αυτό. Ο κύριος Μπόνι πρώτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστούμε κύριε Διευθυντά για αυτήν την ε, επισκόπηση τόσο καλά διαρθρωμένη με ενδελεχή ανάλυση αυτών των τόσο σοβαρών πληροφοριών. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυτό το είδους της ε, παρουσιάσεις εδώ διότι χρειαζόμαστε αυτού του είδους την ενημέρωση για να προετοιμάσουμε τις πολιτικές μας δράσεις. Είναι σημαντικό να είμαστε όλοι ενημερωμένοι για τα νέα ναρκωτικά. Υπάρχουν πολλές νέες τάσεις. Αν συγκρίνουμε το τι συνέβαινε τώρα με το παρελθόν, μετά την επιδημία ηρωίνης στα μέσα της δεκαετίας του 90, βλέπουμε ότι τώρα προκύπτουν προβλήματα από τη χρήση κάναβης ή πρωτίστως από νέες ψυχιενεργές ουσίες, ψυχοτρόπες μάλλον ουσίες. Πιστεύω ότι οι δράσεις μας θα πρέπει να βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία, σε γεγονότα και όχι σε ιδεολογικές σκέψεις. Ως εισηγητής της πρότασης για ένα κανονισμό για τις νέες ψυχοτρόπες ουσίες, ενδιαφέρθηκα ιδιαίτερος για τα πορίσματά σας για τις ουσίες αυτές και πώς σημειώνουν τις τάσεις προσφοράς και ζήτησης. Αφού λοιπόν ανέγνωσα την έκθεσή σας, Πιστεύω ότι μια ισχυρότερη κοινή απόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το φαινόμενο είναι απαραίτητη. Αυτό το κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του το περασμένο έτος και περιμένουμε το Συμβούλιο. Ανησυχώ λίγο που το Συμβούλιο χρειάζεται τόσο πολύ χρόνο και ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε ένα κείμενο που θα προβλέψει αποτελεσματικές και ταχείες διαδικασίες που θα μας επιτρέψουν να καταπολεμήσουμε μαζί αυτό το φαινόμενο. Και χάρη στη δράση του οργανισμού σας και χάρη στη δράση των καταμελών. Δεν έχουμε χρόνο. Παραμένοντας σε διαδικαστικές ε, διαφιλονικίες και παρανοήσεις. Είναι σαφέ από την έκθεσή σας ότι η χρήση αυτών των ουσιών, των νέων ψυχοτρόπων ουσιών, αυξάνεται. Πολύ συχνά προκαλεί προβλήματα στην υγεία και θανάτους. Και οι ουσίε αυτές, όπως κατάλαβα, έχουν να κάνουν με έλλειψη ενημέρωση για τη χρήση τους και των ε, τρόπων αντίδρασης. Είναι τόσες πολλές οι νέες αυτές ουσίες που προκύπτουν διαρκώς, που πολύ συχνά δεν ξέρουμε πώς να συμβάλλουμε από την πλευρά των ε, διοκτικών αρχών για να καταπολεμηθεί η χρήση τους. Διαπιστώνεται ότι πέρα από το ρυθμιστικό και το σκέλος της εκπαίδευσης είναι σημαντικό για την καταπολέμηση της χρήσης. Χρειαζόμαστε πολύ καλύτερα προετοιμασμένους υπευθύνου των διοκτικών αρχών. Και πρέπει να υπάρχει και ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις δράσεις μας. Η έκθεσή σας δείχνει πόσα λίγα ξέρουμε για τις ουσίες αυτές και τις τάσεις που επικρατούν ως προς τη χρήση τους. Σε ορισμένα μέρη, οι νέες ψυχοτρόπες ουσίες δεν καλύπτονται από μελέτες για το τι συμβαίνει ένα κράτος μέλος. Κατά τη συζήτηση λοιπόν για τον κανονισμό θα πρέπει να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να συμβάλλουν στις δικές σας προσπάθειες για να συγκεντρώσουμε περισσότερες γνώσεις περί του θέματος. Και εν τέλει να επαναλάβω ότι χρόνο δεν έχουμε. Χρειαζόμαστε αυτόν τον κανονισμό για να καταλάβουμε καλύτερα το όλο πρόβλημα. Επίσης, το πρόβλημα αυτό έχει να κάνει και με την κάναβη. 20 εκατομμύρια άνθρωποι είναι χρήστε στην Ευρώπη. Από προσωπικής σκοπιάς έχω ένα νέο πρόβλημα στην οικογένειά μου. Ένας από τους, ξα... μία από τις ξαδέλφες μου έχει εξάρτηση από την κάναβη. Το ζω στην οικογένειά μου. Έχουμε λοιπόν ε, πρόβλημα με την κάναβη. Χρειαζόμαστε αποδεκτικά στοιχεία, πληροφορίες και γνώση για να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο. Σας ευχαριστούμε κύριε Μπόνη για αυτές τις παρατηρήσεις και την προσωπική σας μαρτυρία. Γίνονται όλα πολύ πιο ρεαλιστικά έτσι. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Γκέτ για την παρουσίασή σας. Δεν νομίζω ότι κάνατε λόγο για την πώληση και διάδοση του ΚΑΠΤΑ που είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα σε, αυτές τις, ε, σε κάποιες κοινότητες. Και το θέμα του, της ηλικιακής εικόνας και σύνθεσης των χρηστών στην Ευρώπη. Αν έχουν υπάρξει κάποιες αλλαγές σχετικά με την ηλικία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η Μόνικα παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίως μια ερώτηση θα είχα σε δύο θέματα. Πρώτον, είχαμε κατά το παρελθόν σε σχέση με τις προπομπές ουσίες στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μια σε βάθος συζήτηση αν πρέπει να πιστοποιούνται ή αν πρέπει να μπορούν να ειχνηλατούνται, να ανοιχνεύονται, ποια πορεία ακολουθούνται, ποιος πολίτη σε ποιον ποια ποσότητα παράγεται και παρόμοια θέματα, ώστε και η παραγωγή και οι οδοί να μπορούν να ιχνηλατούνται. Αυτό όμως ισχύει μόνο για ουσίες που από τρίτες χώρες εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει άποψη ότι ένας τέτοιος έλεγχος και εξέταση επίσης για τις διαφορετικές ουσίες και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν αναγκαίο να γίνει διότι ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής διεξάγεται στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερο, το θέμα για, το, για την κάναβη. Είπατε ότι 60.000 άνθρωποι βρίσκονται σε θεραπεία, πηγαίνουν σε θεραπεία. Αυτοί είναι εκείνοι που ε, σε χρονική διάρκεια καταναλώνουν κάναβη είναι κάποια ας το πω έτσι ε, ολιστήματα ή λάθη κατά την χρήση κανάβεως που οδηγούν σε αυτή τη θεραπεία ή και κάποιες άλλες ουσίες. Έχετε κάποια ιδέα πώς ε, συναπαρτίζεται αυτός ο αριθμός των 60.000 που βρίσκονται σε θεραπεία. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστούμε Μόνικα. Και τώρα να επιστρέψουμε στον κύριο Γκέτς, αφού πήραν το λόγο οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα απαντήσω και στους τρεις με τη σειρά. Κύριε Μπόνη, είπατε ότι υπάρχει ανάγκη για ρύθμιση του φαινομένου, για να αναλάβουμε δράση ρυθμιστική. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω χρειάζεται νομική βάση για τις νέες ψυχοτρόπες ουσίες, διότι όσα έχουμε τώρα βασίζονται στην τελευταία νομοθεσία του 2005, με προηγούμενη νομική βάση από το 1997. Είναι λοιπόν απερχιωμένα όλα αυτά σε σχέση με τα σημερινά φαινόμενα. Από τη δική μου τη σκοπιά, από τη σκοπιά του ε, οργανισμού, του κέντρου μας, έχουμε δύο ε, σημαντικά πράγματα να πούμε. Ότι πρέπει να υπάρξει μια σταθεροποίηση και επίση ένα σύστημα γύρι προειδοποίηση ενδεχομένω. Αυτέ είναι οι προτεραιότητε του κέντρου μα. Σίγουρα η Επιτροπή έχει άλλε προτεραιότητε όπω η νομική βάση και το καθεξή. Η κάναβη τώρα. Είναι μια ουσία που συζητείται πάρα πολύ σήμερα. Διότι υπάρχουν ε, θέματα κανονιστικών ε, ρυθμίσεων ή της νομιμοποίησης ε, στι ΗΠΑ και αλλού. Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι ότι έχει γίνει πιο επικίνδυνη ουσία η κάναβη από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Όταν ήμουν 16, τη δεκαετία του 60 και του 70, ήταν απλό να καπνίσει κανείς ένα τσιγάρο κάναβης με τους φίλους του, μια στις τόσες. Σήμερα όμως είναι διαφορετική η ουσία. Είναι πολύ ψηλότερες οι είναι πολύ υψηλότερη η περιεκτικότητα σε THC ε, για λόγω των λοιπασμάτων που χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια της κάναβης και ούτω καθεξής ή όσων προέρχονται ε, από το Μαρόκο και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν, να μην ξεχνάμε ότι όσοι μιλάνε για διευθέτηση του προβλήματος της κάναβης με διαφορετικούς κανονισμούς και κανόνες, γνωρίζουν πολύ καλά αυτό το πρόβλημα. Δεν ανέφερα το κάτι που είναι συγκεκριμένο πρόβλημα για ανθρώπους από ορισμένες κοινότητες, όπως ε, ανθρώπους που προέρχονται από τον Τζιμπουτί, τη Σομαλία και το καθεξής. Το Ενωμένο Βασίλειο πέρσι έλαβε μέτρα για το θέμα αυτό. Νομίζω και κάποιες σκανδιναβικές χώρες, αλλά πρέπει να ομολογήσω, έχω ένα συνάδελφο που είναι ειδικό για τα θέματα αυτά. Ε, για την ουσία αυτή. Εγώ δεν τα ξέρω τόσο καλά. Για τι ε, συνθετικές ουσίες τώρα, τα καφεϊνοειδή λόγω χάρη, έχουν παρόμοιες συνέπειες και επιπτώσει με την κατανάλωση κάτι. Είναι συνθετικά και δεν χρησιμοποιούνται από αυτού για του οποίου η χρήση ΚΑΤ είναι σχεδόν ε, πολιτιστικό θέμα, παρά, θέμα παράδοση. Ιδίω ε, για όσου προέρχονται από χώρε τη Ανατολική Αφρική. Το πιο σημαντικό ε, από όλα αυτά είναι το τι γίνεται με τους χρήστες ηρωίνης. Είναι όλο και χαμηλότερης ηλικίας αλλά έχουμε φτάσει σε ένα μέσο όρο ηλικίας ε, που έχει αυξηθεί κατά πέντε χρόνια πλέον. Υπάρχει ανάγκη να περιθάλψουμε αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχουν ήδη σε κάποιες χώρες ιδέες για οίκους ευγυρίας για χρήστες ηρωίνης. Δεν ξέρουμε πώς αυτό μπορεί να λειτουργήσει. Δυστυχώ δεν ανήκουν αυτές οι ουσίες που αναφέρατε στη δική μου εντολή. Πρόκειται για εντολή τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν θέλω να αναμειχθώ ιδιαίτερα. Όμω, οι αριθμοί είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην έκθεσή μας η σελίδα 36 της αγγλικής ε, έκδοσης έχουμε πληροφορίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά Γενικά μπορούμε να πούμε ότι φυσικά ενδιαφερόμαστε οι προπομπές ουσίες να μπορούν να ελέγχονται όσο το δυνατόν περισσότερο, αλλά πρέπει να δούμε ότι πολλές από αυτές τις ουσίες χρειάζονται, τις χρησιμοποιεί ε, η βιομηχανία. Και τίθεται το ερώτημα, πώς θα είναι κάτι τέτοιο εφικτό. Είναι όμω ένα σημείο στο οποίο δεν θα ήθελα να αναμειχθώ με δικέ μου παρατηρήσει. Δεν θα το εκτιμούσε η Επιτροπή αν το έκανα. Οι 60.000 τώρα υποθεραπεία αυτά τα άτομα. Είναι άτομα που για πρώτη φορά μεταβαίνουν προς θεραπεία. Αναφέρουμε αυτό τον αριθμό, είναι η πρώτη φορά που μεταβαίνουν προς θεραπεία. Οι επιστρέφοντες και άλλοι δεν συμπεριλαμβάνονται. Νομίζω ένα τρίτο θα πρέπει να είναι που ε, αποστέλλονται από το δικαστικό σύστημα, από τα δικαστικά κυκλώματα εκεί. Θεραπεία είναι απόφαση για παράδειγμα δικαστών. Λέει ένας δικαστής, εσύ θα πας ως κατηγορούμενος τώρα σε θεραπεία. Πρέπει να το δούμε, δεν είναι όλοι εθελοντικά υποθεραπεία λοιπόν. Αυτά ήταν ε, αυτά τα οποία μπορούσα να πω για τα πολύ συγκεκριμένα ερωτήματά σας και όπως προανέφερα στην αρχή το κάνουμε αυτό τώρα 20 χρόνια όχι εγώ αλλά η υπηρεσία μας επιτελεί αυτό το έργο επί 20 χρόνια. Έχουμε μια τελείως διαφορετική κατάσταση από ό,τι πριν από 20 χρόνια. Η κατάσταση δεν είναι, δεν θα έλεγα πιο προβληματική, αλλά είναι πολύ πιο σύνθετη και περίπλοκη. Και αυτό καθιστά όλο και περισσότερο δυσχερές να ανοιχνευθούν τα πάντα και να έχουμε όλες τις πληροφορίες όπως απαιτείται. Θέλω όμως να ευχαριστήσω όλους τους εταίρους που εμπλέκονται σε αυτό το έργο κράτη-μέλη και τα εθνικά εστιακά σημεία focal points αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι καθημερινός εταίρος σε αυτό το έργο και από της τεχνικής πλευράς, όχι πάντα από πλευράς προϋπολογισμού, εξαιρετικός εταίρος. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και να πω ότι σε τακτά διαστήματα συμμετέχουμε στην οριζόντια εγκάρσια ε, ομάδα της Επιτροπής. Θέλω να ευχαριστήσω και την Ευρωβουλή ιδιαίτερα την Επιτροπή τη δική σας για την υποστήριξη που μας προσφέρατε όλα αυτά τα έτη μέχρι σήμερα. Και ίσως είναι η τελευταία φορά που παρίσταμε εδώ, δεν το γνωρίζω. Ε, έληξε, εξέπνευσε ήδη η εντολή, η θητεία μου, άρα είναι δύσκολο να βρεθεί διάδοχος. Θα παραμείνω μέχρι την εξέβρεση επόμενου διευθυντή. Ίσως δηλαδή μέχρι τους πρώτους δύο μήνες του επόμενου έτους. Ευχαριστώ. Um, Ευχαριστούμε. Θα δώσουμε το λόγο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αναφέρατε σύντομα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λίγα λόγια να ευχαριστήσω τον κύριο Γκέτ, τον Διευθυντή του Κέντρου, για αυτή την εξαιρετική παρουσίαση τη έκθεσή του. Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο για την Αντιμετώπιση του Φαινομένου Κατανάλωση Ναρκωτικών, όπω καταγράφεται στη στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση κατά των Ναρκωτικών, βασίζεται πάρα πολύ ε, στα αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώνουμε. Γι' αυτό είμαστε ευγνώμονες προς το κέντρο που ετοιμάζουν μια τέτοια έκθεση τόσο σημαντική για τους σχεδιαστές πολιτικής. Το κέντρο είναι πρότυπο όχι μόνο για τους άλλους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και ο ρόλος του Διευθυντή υπήρξε καθοριστικός στη λειτουργία του κέντρου. για τις ε, νέες συνθετικές ουσίες, ε, όντως ανάγεται η νομική βάση στο 2005, δεν μπορούμε να καλύψουμε έτσι τις νέες ψυχοτρόπες ουσίες που χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι η παραγωγή ναρκωτικών και οι έμποροι φέρνουν την παραγωγή εδώ, όπου η αγορά είναι πιο πρόσφορη. Τα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον αυτό, όμω δυστυχώ επί ηλεκτρονική προεδρία δεν μπορούσαμε να επιτελέσουμε πρόοδο στο Συμβούλιο. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε τώρα με την επόμενη προεδρία. Και τώρα δύο λόγια για τη διεθνή διάσταση. Και εκεί καλωσορίζα όσα υπόθηκαν από τον κύριο Γκέτ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μιλά με ενιαία φωνή στο διεθνέ προσκήνιο. Και υπολογίζουμε στη δράση του Επιτρόπου Αβραμόπουλου, ο οποίος συνεργάζεται και θα συνεργαστεί με την Προεδρία για να ετοιμάσουμε μια ισχυρή θέση ε, του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο και της ανάλογης επιτροπής του ΟΗΕ που θα συνέλθει την ε, επόμενη χρονιά. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ κύριε Γκέτς για τη δουλειά σας. Δεν είναι η τελευταία φορά που θα σας δούμε εδώ. αλλά με την παρέμβαση των συγκητών μας, των συνεισηγητών μας και των ε, σκιωδών συγκητών, καταλαβαίνετε ότι και οι δικές γνώσεις μας ενδιαφέρουν και το ενδιαφέρον μας παραμένει αμύωτο για τα θέματα αυτά. Ελπίζουμε να συνεχίσετε και εσείς τις προσπάθειές σας και σας ευχαριστούμε. Θα σας ξαναδούμε. Ευχαριστούμε. Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, προχωρούμε τώρα στην έκθεση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο για τη λειτουργία του χώρου Σέγγεν. Είναι μια έκθεση η οποία δημοσιεύεται ε, κάθε δύο χρόνια. Να σας πω ότι την περασμένη Κυριακή είχαμε μια επέτειο που θα ήθελα να αναφέρω. Είναι η επέτειος της σύναψης της Συμφωνίας Σέγγεν, η οποία όπως γνωρίζουμε όλοι ε, υπογράφει στις 14 Ιουνίου του 1985 και νομίζω ότι πρέπει να αποτίσουμε φόρο τιμή στους ανθρώπους που είχαν το θάρρος να κάνουν τότε ένα τέτοιο βήμα. Η εύρεθμη λειτουργία του χώρου Σέγγεν είναι κάτι πολύ σημαντικό για εμάς και καλωσορίζουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία θα μας υποβάλει και θα μας παρουσιάσει την διετή της έκθεση για τη λειτουργία του χώρου Σέγγεν. Θα ε, πρέπει να πω ότι το Σέγγεν, ο χώρος Σέγγεν είναι ακόμα πιο σημαντικό σήμερα από τη στιγμή που ε, έχουμε διάφορα ε, πρακτικά θέματα εφαρμογής της συμφωνίας. Είναι ο κύριος Ντεκόιστερ εδώ. Ναι, έχετε το λόγο. Θα μας κάνετε μια σύντομη παρουσίαση και μετά θα υπάρξει συζήτηση. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Όπως γνωρίζετε, κάθε έξι μήνες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει δυο φορές το χρόνο την έκθεση για το χώρο Σέγγεν. Είναι η έβδομη λοιπόν έκθεση ε, που έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29 ε, Μαΐου. Ε, Δις ετησίως λοιπόν δημοσιεύεται η έκθεση για τη λειτουργία του χώρου Σέγγεν, η οποία ε, καλύπτει όλες τις σχετικές πτυχές του θέματος αυτού. Η έβδομη έκθεση αφορά την περίοδο 1η Νοεμβρίου 2014 μέχρι 30 Απριλίου 2015, αυτό το εξάμεινο. Η περίοδος αναφοράς χαρακτηρίστηκε κυρίως και πάνω απ' όλα από τα τραγικά γεγονότα στη Μεσόγειο, από την πίεση στα ουγγροσερβικά σύνορα και από τις από απειλές των ξένων μαχητών της τρομοκρατίας. Θα ήθελα λοιπόν στην παρέμβασή μου να επικεντρωθώ σε αυτά τα τρία ζητήματα παρόλο που η έκθεση στη γραπτή της μορφή αναφέρεται σε πλειάδα άλλων ζητημάτων που σχετίζονται με την εύρυθμη λειτουργία του χώρου Σέγγεν. Ως προς την παράτυπη μετανάστευση. Τρεις είναι οι βασικές οδοί μέσω των οποίων λαμβάνει η χώρα η παράτυπη μετανάστευση προς την Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια της περίοδου αναφοράς του εξαμήνου αυτού, ο υψηλότερος αριθμός ε, προσεγγίσεων ήταν από την οδό των Δυτικών Βαλκανίων, περισσότερες από 62.000 προσεγγίσεις, apprehensions. Όμως αυτό το πρόβλημα έχει αποκατασταθεί λόγω των παρεμβάσεων και η κατάσταση μπορεί να ε, σταθεροποιηθεί και να λυθεί. Από 60.000 το ε, Φεβρουάριο είχαμε 15.000 το Μάρτιο και 7.000 τον Απρίλιο. Οι κοσοβάροι που ανοιχνεύτηκαν στα ουγγροσερβικά σύνορα ήταν περίπου 12.000 το Φεβρουάριο και λιγότεροι από 3.000 τον Απρίλιο. 300 ε, ε, τον Απρίλιο, με συγχωρείτε. Και όλα αυτά οφείλονται στα μέτρα που έχουν ληφθεί. Ε, είχαμε τη στήριξη της Frontex στις Ουγγρικές Αρχές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει έναν εντατικό διάλογο με τη Σερβία και το Κοσφοπέδιο, ο οποίος οδήγησε σε καλύτερη συνεργασία μεταξύ των αρχών αυτών των χωρών. Επομένως, η επισκόπηση αυτών των μέτρων ε, αναλυτικά παρουσιάζεται στην έκθεση αυτή καθ' αυτή. Έρχομαι τώρα στην κατάσταση στην κεντρική Μεσόγειο, η οποία αποτελεί και την πιο σημαντική πρόκληση για εμάς μία από τις πιο σημαντικές. Κατά τη διάρκεια της περίοδου αναφοράς είχαμε 42.000 προσεγγίσεις, apprehensions, ενώ ε, το σώσιμο της ανθρώπινης ζωής είναι η απόλυτη προτεραιότητα για όλα τα θεσμικά όργανα, η διάσωση της ανθρώπινης ζωής και για το Κοινοβούλιο και για το Συμβούλιο και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό το στοιχείο αποτελεί μέρος της έκθεσης Schengen, όμως οι προκλήσεις δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με τα εργαλεία που που διατίθενται βάσει της συνεργασίας Σέγγεν. Χρειάζονται και άλλα διότι οι λανθάνουσες αιτίε είναι εκτός του πλαισίου Σέγγεν. Άρα το κεκτημένο Σέγγεν δεν μπορεί να μας οδηγήσει σε κατάλληλη δράση έτσι ώστε να τελειώσουμε με αυτά τα προβλήματα. Βεβαίως τα μέτρα Σέγγεν μπορούν να προσφέρουν κάποιες λύσεις και αναφέρομαι κυρίως στη συνεργασία μέσω της Frontex με τα κράτη-μέλη για κοινέ επιχειρήσεις και δράσεις όπως είναι ο Ποσειδώνας. Έχετε ήδη λάβει πλήρη ενημέρωση και πληροφορίες για την εφαρμογή αυτών των αποκοινού δράσεων, joint operations. Επομένως, αναλάβαμε κάποια δράση, χρησιμοποιήσαμε κάποια εργαλεία Σέγγεν και τα χρειαζόμαστε όλα αυτά, αλλά χρειαζόμαστε και άλλα μέτρα και άλλου είδους δράσεις. Και εδώ εννοώ την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τη Μετανάστευση και το πακέτο εφαρμογής των σχετικών κινημένων, έτσι όπως το έχει υιοθετήσει πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επομένως, η Κεντρική Μεσόγειος αποτελεί και μία από τις πιο σοβαρές προκλήσεις σήμερα. Να μην λησμονούμε όμως ότι υπάρχουν και άλλες μεταναστευτικές δίωδοι ή οδοί και ε, πρέπει να υπάρχει επαρκής επιτήρηση από την άλλη πλευρά των εξωτερικών συνόρων. Οι διακινητές πολύ γρήγορα προσαρμόζουν τον τρόπο λειτουργίας τους. Για παράδειγμα στην οδό της Ανατολικής Μεσογείου, αυτό, αυτή ήταν η κύρια οδός που χρησιμοποιήθηκε το Μάρτιο και έφτασε στα επίπεδα σχεδόν της Κεντρικής Μεσογείου από πλευράς προσεγγίσεων, apprehensions. Όμως, ενώ στην Κεντρική Μεσόγειο. Η μεγαλύτερη σημασία δίδεται στη διάσωση της ανθρώπινης ζωής γιατί η, τελικά η επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων καταλήγει σε επιχείρηση διάσωσης ανθρώπινης ζωής ανθρωπιστικής. Αυτό ενδεχομένως δεν ισχύει στις άλλες πλευρές της Μεσογείου. Ένα δεύτερο που θα πρέπει να αναφέρω είναι η λειτουργία του νέου μηχανισμού αξιολόγησης Σέγγεν, ο οποίος έγινε πλήρως εφαρμόσιμος το Νοέμβριο της περασμένης χρονιάς. Οι πρώτες αξιολογήσεις έγιναν στην Αυστρία και στο Βέλγιο και οφείλω να πω ότι η συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών ήταν εξαιρετική και η πρώτη έκθεση για την αξιολόγηση π.χ. της Αυστρίας υποβλήθηκε την περασμένη Παρασκευή στην Επιτροπή Σέγγεν η οποία θα εκδώσει γνώμοδότηση για αυτά τα σχέδια εκθέσεων. Όπως γνωρίζετε προβλέπεται στην απόφαση του Συμβουλίου που θεσπίζει ένα νέο μηχανισμό αξιολόγησης και μέσα σε αυτή την απόφαση προβλέπεται ότι οι εκθέσεις αξιολόγησης θα διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχει τώρα το θέμα των ξένων μαχητών τρομοκρατίας για τους οποίους έχουν υποβληθεί εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως γνωρίζετε, το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο επιτρέπει τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων και δεν υπάρχει ανάγκη να αλλάξει π.χ. ο κώδικας των συνόρων βάσει του Σέγγεν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάστηκε να υιοθετήσει συστάσεις για να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να στοχοθετήσουν καλύτερα τους ελέγχους στα άτομα, στα πρόσωπα που αξιοποιούν την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των Ευρωπαίων πολιτών. Γνωρίζετε ότι συστηματικός έλεγχος αυτών των προσώπων δεν επιτρέπεται σε γενικές γραμμές από τον κώδικα των συνόρων, όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε μία ερμηνεία που επιτρέπει ελέγχους με καλύτερη στόχο προσήλωση, με καλύτερη στόχο θέτηση και δηλώνει ότι με βάση την ανάλυση των κινδύνων εσωτερικής ασφάλειας και με βάση την ανάλυση των τάσεων που μπορεί να πλήξουν την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων μπορούν να γίνονται συστηματικοί έλεγχοι στα λόγω πρόσωπα που είναι δικαιούχοι της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τη στιγμή που τα πρόσωπα αυτά παρουσιάζουν κριτήρια που εντάσσονται στην αξιολόγηση κινδύνου. Και έχουμε ήδη ε, δει ότι κράτη-μέλη κάνουν αυτή τη σύσταση και υπάρχουν τέτοιοι έλεγχοι. Και όσον αφορά τα ταξιδιωτικά έγγραφα εκείνων που υποφελούνται από την ελεύθερη κυκλοφορία και έχουμε και ελέγχους ατόμων που αφορούν αυτούς τους, ε, ε, αυτά τα άτομα. Όπως είπα Πρόεδρε, υπάρχουν και πολλά άλλα θέματα τα οποία καλύπτονται όπως για παράδειγμα το θέμα της Eurosur οι εξελίξεις όσον αφορά θεωρήσεις διαβατηρίων. Θα ήθελα όμως να επιστήσω την προσοχή σας και σε μια άλλη πτυχή που είναι όπως εσείς επισημαίνετε, επισημάνατε εισαγωγικά η επετηρίδα της υπογραφής της Συμφωνίας Σέγγεν. Και σε σχέση με αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί την πλήρη υποστήριξή της προς την Βουλγαρία και Ρουμανία να ενταχθούν στον χώρο Σέγγεν. Δεύτερο στοιχείο μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα έπρεπε επίσης να αναφέρω ότι η Κροατία ίδια δύο μήνες πριν επίσημα δήλωσε ότι είναι πρόθυμη να αξιολογηθεί από πλευρά του Σέγγεν. Θεωρεί λοιπόν ότι θα μπορούσε να περάσει τη δοκιμασία, το τεστ αυτό όσον αφορά την ένταξη της στο χώρο Σέγγεν. Μπορώ να σας ενημερώσω ότι ήδη προσαρμόζουμε το πολιτές πρόγραμμα αξιολόγησης ώστε να έχουμε και τις επισκέψεις που θα πρέπει να διεξαχθούν αρχές του 2016 στην Κροατία σχετικά. Όπως γνωρίζετε η έκθεση, όπως ε, γνωρίζετε Πρόεδρε, είναι μια απεικόνηση, ένα στιγμιότυπο το οποίο απεικονίζουμε. Αυτές οι ε, θεωρήσεις διαβατηρίων ε, αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, άρχισαν να ισχύουν προσωρινά και σε σχέση με την συζήτηση στην Επιτροπή σας στις 15 ε, Ιουλίου. Άλλα επίσης θέματα έχουν εξελιχθεί και αυτά παράλληλα και φυσικά το, πιο σημαντικό ε, εξέλιξη <clears throat> συνέβη μετά την περίοδο αυτή ε, για την έκθεση που είναι η, τα θέματα μετανάστευσης και η συνολική σφαιρική προσέγγιση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θέματα μετανάστευσης ώστε να τύχουν καλύτερης διαχείρισης. Αυτή η έκθεση σε αντίθεση με άλλες προηγούμενες εκθέσεις στα συμπεράσματά της ε, δεν θέτει ερωτήματα προς πολιτική συζήτηση. Το πραγματικό ζήτημα το οποίο εδώ βρίσκεται υπό διακύβευση είναι η καλύτερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και η αντίδραση στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Μεσόγειο. Αυτή η συζήτηση διεξάγεται ήδη και την παρακολουθείτε και εσείς και το Συμβούλιο. Δεν διατυπώσαμε κάποια άλλα θέματα τα οποία θα έπρεπε να συζητηθούν συγκεκριμένα μέσα στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης. Αυτά είχα να πω Πρόεδρε. Είμαι πρόθυμος και στη διάθεσή σας να απαντήσω σε παρατηρήσεις και ερωτήσεις. Thank Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Δικαστήριο. Θα σημειώσετε, συνάδελφοι, ότι παρόλο που ήταν σύντομη η παρουσίαση, περιείχε πολλά θέματα προς συζήτηση. Η συμφωνία του Σέγγεν είναι το βασικό θέμα, όμως αγγίζει πολλές άλλες εκθέσεις και θέματα που μας απασχολούν. Είναι πολλά αυτά που θα μπορούσατε να σχολιάσετε report migration other areas where we can discuss these points. So... Είναι πολλοί λοιπόν οι τομείς που άπτονται αυτού του θέματος και θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Σας ευχαριστούμε για αυτή τη λεπτομερή και διεξοδική ε, παρουσίαση κύριε Κέστερ. Έχω ένα μακροσκελή κατάλογο μιλητών λοιπόν μετά από αυτή την παρουσίαση. Ξεκινώ με τον κύριο Κοέλιου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, συνάδελφοι, να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την παρουσίαση αυτή τη έκθεσης, αλλά πρέπει να πω ότι λυπούμε που δεν μπορούμε να έχουμε καλύτερο έλεγχο των θεμάτων αυτών, γιατί ο χώρο Σέγγεν και το κεκτημένο Σέγγεν έχουν δεχτεί πίεση, όπως είπε και ο κ. Κέστερ ήδη έχουν να κάνουν με τον πυρήνα των ε, ενδιαφερόντων των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά με την ανάδυση τρομοκρατίας και εξτρεμιστών, βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί στενότερα τα θέματα αυτά. Ελπίζω, Πρόεδρε, στην επόμενη τουλάχιστον έκθεση να έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μα. Το Σέγγεν είναι ζωτική σημασία για την Ευρώπη των πολιτών και θα πρέπει να είναι μία από τι ύψιστε προτεραιότητε αυτή τη Επιτροπή. Η έκθεση αυτή ήταν όντω καλή και παρόλα αυτά θα πρέπει να περιέχει λεπτομερέστερα στοιχεία. Να σταθώ σε τρία σημεία και να θέσω ερωτήσει προ τον κύριο Ντεκέστερ. Πρώτα απ' όλα, η Επιτροπή δεν δείχνει πώ θα υπάρχει καλύτερη αστυνομική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με τη Σερβία ώστε να μειωθεί η παράτυπη μετανάστευση μεταξύ Σερβίας και Ουγγαρίας και Κωσυφοπεδίου. Δεύτερον, ε, η έκθεση αυτή από 1η Νοεμβρίου 2004 μέχρι σήμερα καλύπτει το χρονικό διάστημα, όμως αναφέρεται σε 13 επιχειρήσεις που ξεκίνησαν ε, ε, ε, με ακρίβεια την 1η Νοεμβρίου. Και τα στοιχεία δεν είναι αρκετά για να καταλήξουμε σε πολιτικές θεωρήσεις σε πολιτικέ παρατηρήσει. Το μέλλον θα είναι καλύτερα να ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιο αντικειμενική στην εξέταση του θέματο αυτού. Για, και Μιλήσαμε για τεπλασιασμό της χρηματοδότησης των ε, αποστολών αυτών. Η Επιτροπή μας ε, χθες ζήτησε μία τοποθέτηση για τις περικοπές που έχουν γίνει στις διάφορες λειτουργίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει να σχολιάσει γι' αυτό και επίσης η έκθεση λέει ότι αυτό το μήνα θα υπάρξει μία πρώτη έκθεση για τις δευτερογενείς μετακινήσεις. Υπάρχει καμία πρόπτικη για το πότε θα έχουμε κι εμείς πρόσβαση στα στοιχεία αυτά. Και τέλος, Πρόεδρε, Και τώρα μία, ε, ένα σχόλιο για την τολμηρή κίνηση της Επιτροπής να ε, απαιτήσει στοιχεία για την οδηγία της επιστροφής. Η Γαλλία και η Ιταλία έχουν υποβάλει διαδικασία με έχουν προσφύγει με παραβάση για το θέματα αυτά μη μετακίνησης, αλλά και για τη Ρωμανία και τη Βουλγαρία που έχουν συμμορφωθεί πλήρω με τα αυστηρά κριτήρια της οδηγίας αυτής. Δεν θα πρέπει να πιέσουμε το Συμβούλιο για να προχωρήσει στο θέμα αυτό. Και τέλο. εξίσου σημαντικό, οι παρατηρήσει για τον νέο μηχανισμό αξιολόγηση του Σέγγεν. Όπω ε, ο κανονισμό αυτό μόλι τέθηκε σε ισχύ, είναι ζωτική σημασία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τον αξιοποιεί πλήρω. Εξαρτάται πλήρω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη προπολή σε αυτόν τον πλήρω ευρωπαϊκό μηχανισμό. Ε, με όλα τα νέα μέσα πρέπει να ενισχύσουμε την αμοιβή συνεργασία μεταξύ των κρατομελών και πρέπει να βεβαιωθούμε ότι έχουμε ε, ισχυρά και προστατευμένα σύνορα. Είναι ζωτική σημασία να είμαστε βέβαιοι ότι τα κράτη-μέλη συμμορφώνονται με, τον, ε, με την ουσία του κεκτημένου Σέγγεν. Όλα αυτά μπορούμε να πετύχουμε μόνο μέσω ενό αποτελεσματικού μηχανισμού αξιολόγηση που βρίσκεται στα χέρια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ερώτησή μου είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τα μέσα να επιτελέσει αυτά τα νέα καθήκοντα. Και θα ε, υποβάλω και κάποιε ερωτήσει, αν χρειαστεί. Ελπίζω, Πρόεδρε, ότι κάλυψα τα ζωτικότερα σημεία. Ευχαριστούμε, κύριε Κοέλιο. Είναι όντω πάρα πολλά αυτά που θα μπορούσαμε να πούμε. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα του Σέγγεν που είναι σημαντικά, σωστά τα επισημάνατε και ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα με το οποίο θα προκύπτουν θα τα συμπεριλαμβάνουμε και στην ημερήσια διάταξη. Αυτό το θέμα περιλήφθη για επαιτειακούς λόγους. Όντω, σε επόμενη φάση θα προβλέψουμε μια μακροσκελέστερη συζήτηση και θα καλύψουμε το θέμα αυτό του Σέγγεν. Αυτό που επισημάνατε εσεί είναι ε, το τι σκέφτεται ένα ειδικό επί του θέματος για τα θέματα του Σέγγεν. Συνάδελφοι όμω πρέπει λίγο να βιαστούμε. Πολύ σύντομα θα έχουμε τα συμπεράσματα τη Λεπτονικής Προεδρία. Θα σα έλεγα λοιπόν επειδή το σημείο αυτό έχει επαιτειακή και συμβολική σημασία, να προσπαθήσετε να περιοριστείτε στο ένα λεπτό στα σχόλιά σας ε, θα ακούσουμε την κυρία Σπινέλη, Ντούντα, Αρχεντίνη και ούτω καθεξής. Παρακαλώ περιοριστείτε σε ένα λεπτό για να προλάβουμε. Θα έχουμε και άλλο σημείο για το, για το Σέγγεν, πολύ σύντομα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και για την αναφορά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνάδελφοι, 8 χρόνια μετά την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποφέρει από, από πολλά μέτρα και σταθμά η χώρα μας. Υπάρχουν πολιτικοί σε κράτη-μέλη που διασπείρουν λανθασμένες πληροφορίες όσον αφορά τη Βουλγαρία. Ιδιωτελώς το πιο εξόφθαλμο παράδειγμα είναι ότι η Βουλγαρία βρίσκεται εκτός χώρου Σέγγεν Πολλοί έλεγχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακάλυψαν, διαπίστωσαν ότι η χώρα μας ανταποκρίνεται σε όλα τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο εισηγητής ο κ. Κάρλος Κοέλιο, τον οποίο ευχαριστώ θερμά για την μακρά υποστήριξη που μας παρήχε, επανειλημμένα ζήτησαν η Βουλγαρία να ενταχθεί στην, στον χώρο Σέγγεν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό γίνεται και στην 7η έκθεση που κατατέθηκε πριν από λίγο είναι καθαρή εισφορέας η Βουλγαρία στην, ε, στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και οι μεθοριακοί φύλακες με επιτυχή τρόπο φυλάσσουν τα σύνορά μας προς την Τουρκία και ο αριθμός των μεταναστών που ε, διασχίζουν αυτά τα σύνορα είναι πολύ μικρότερος από εκείνους ε, που διασχίζουν τη Μεσόγειο και καταλήγουν σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο κύριος Μπόικο Μπορίσοφ, ο Πρωθυπουργός μας, ε, έχει τοποθετηθεί. Πολύ λίγοι διασχίζουν τα σύνορά μας. Παρ' όλα αυτά η Βουλγαρία δεν είναι κράτος μέλος του Σέγγεν και αυτό είναι απαράδεκτο και δεν δείχνει σεβασμό προς τους Βουλγάρους. Καλό τα κράτη-μέλη να αποδείξουν ότι θεωρούν ότι η Βουλγαρία είναι πλήρε μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό μπορεί να αποδειχθεί μόνο αν η χώρα επιτραπεί να γίνει κράτο μέλο τη Σέγγεν. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπερζιά παρακαλώ. Η κυρία Μπερζιά. Ευχαριστώ πρόεδρε. και εγώ θα ήθελα να έχουμε επέτειο του χώρου Σέγγεν και να μπορώ να το γιορτάσω, εάν υπήρχε όμως και ένας χώρος ελεύθερης κυκλοφορίας που να λειτουργεί πραγματικά και να βασίζεται σε σωστές συνθήκες. Ε, και ακόμα λιγότερο δεν μπορώ να θεωρήσω ότι πρέπει να γιορτάσουμε την επέτειο της οικοδόμησης ε, ενός οχυρού Τη Ευρώπη με κλειστά σύνορα. Δυστυχώ αυτό ισχύει όλο και περισσότερο. Βλέπω λοιπόν ότι οι περισσότερες συζητήσει που γίνονται στα κράτη-μέλη για το θέμα αυτό δεν έχουν την σωστή τοποθέτηση. Ε, είναι λίγο κακοπροαίρετε, διότι δεν φαίνεται όταν αμφισβητεί το χώρο Σέγγεν να ξέρουν οι άνθρωποι γιατί μιλάνε, ακόμη και για τα όρια του. Το άλλο στοιχείο που ήθελα να αναφέρω και δεν είναι σφάλμα του της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι ότι έχουμε πρόβλημα ως προς την παρουσίαση των αριθμητικών στοιχείων και το πώς παρουσιάζονται. Ε, δηλαδή πώς αξιοποιούνται ή γίνονται αντικείμενα εκμετάλλευση στα ποσοστά. Ένα παράδειγμα, πολύ σύντομα μας δόθηκε εξήγηση ότι η πίεση στα εξωτερικά σύνορα της Ελλάδας έχει αυξηθεί κατά 100%. Ε, αλήθεια είναι αυτό, αλλά τα ποσοστά μπορεί κανεί να τα ερμηνεύει όπω θέλει. Εξαρτάται από ποια σκοπιά τα βλέπει κανεί σήμερα η μεταναστευτική πίεση είναι περίπου η ίδια για την Ελλάδα και την Ιταλία. Οι αριθμοί λοιπόν είναι περίπου 50.000 σε κάθε χώρα. Η κατάσταση της Ελλάδας δεν είναι σαφώς η ίδια με αυτήν της Ιταλίας. Ε, υπογραμμίζω ότι η Ελλάδα δεν έχει πάρει ούτε ένα ε, λεπτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα λεπτό του ευρώ, για τα θέματα αυτά. Έχουν μπλοκαριστεί όλα για λόγους που δεν θα ε, αναλύσω τώρα, τους γνωρίζετε όλους. Το βρίσκω σκανδαλώδες. Είναι ένα ξεκάθαρο σκάνδαλο. Υπάρχει λοιπόν παραποίηση των στοιχείων αυτών υπάρχει η αξιοποίησή τους για τους σκοπούς που θέλει ο καθένας και θα πρέπει να προσέξουμε να μην δίνουμε επιχειρήματα στις ξενοφοβικές ε, συζητήσεις. Και επειδή είμαι Γαλλίδα, θέλω να σας πω και το εξής κύριε Πρόεδρε, για κάτι που συμβαίνει στη Νίκαια. Εδώ και χρόνια η Γαλλία έχει κλείσει τελείως τα σύνορά της μεταξύ Ιταλίας και ημών. Τι γίνεται λοιπόν, γίνονται έλεγχοι ε, ε, διαζώσει. Ε, ε, αναγκάζουν του ανθρώπου να κατέβουν από τα τρένα εφόσον έχουν ύποπτη όψη. Τα τρένα που έρχονται από την Ιταλία προ την Νίκαια. Αυτό το βρίσκω σκανδαλώδε και θα θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μα ε, κάνει σχόλιο για αυτό που γίνεται εδώ και κάποιε μέρε στη Γαλλία και το οποίο το βρίσκω τελείω απαράδεκτο. Πρόεδρο, ευχαριστούμε κυρία Σπινέλη. Μπάρμπαρα, ξέρω ότι είναι θέμα Σέγγεν, αλλά αν μπορείτε σύντομα τα σχόλιά σα γιατί έχουμε πολύ φορτωμένη ημερήσια διάταξη. Μέχρι τι 10.45, οπότε θα πρέπει λίγο να βιαστείτε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θα μακρηγορήσω. Δεν θα επεκταθώ για τα όσα συμβαίνουν στην ε, Νίκαια και στην Ιταλία. Τα ανέφερε η συνάδελφος. Ξέρουμε τι προκαλούν ε, τα μέτρα του Σέγγεν. Έχω όμως ακόμα δύο ερωτήσεις. Ένα. Για τα κονδύλια που δεν φτάνουν ως την Ελλάδα, το ανέφερε η Μαρή Κριστίν, το βρίσκω σκανδαλώδες αυτό, ιδίως επειδή αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι σχεδόν σε default, σε πτώχευση. Και μία ερώτηση. Είπε ότι υπάρχει μια κοινή ερμηνεία των ξένων μαχητών ο εισηγητής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό το σύστημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βασίζεται σε εγκύκλιο. Είναι μια εγκύκλιο που το Κοινοβούλιο δεν την γνωρίζει. Πότε δημοσιοποιήθηκε και πώς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μπάρμπαρα, ευχαριστώ που ήσουν σύντομοι. Η κυρία Σαρχεντίνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ήθελα πράγματι να ερωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα μπορούσαν πιο εξειδικευμένα να πούν για αυτά τα οποία είδαμε αυτό το Σαββατοκύριακο στα σύνορα Βεντιμίλια, Μαντών. Ξέρω ότι είναι εκτό ε, αυτή τη έκθεση, αλλά συνέβη αυτό το Σαββατοκύριακο και θα ήθελα κάποιε πληροφορίες. Θα ήθελα να ζητήσω από τον πρόεδρο, εσά, Κλοντ Μωράης, αν θα μπορούσαμε να αποστείλουμε μια επιστολή προς την Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επίσημα ερωτώντας σε ποιου κανονισμούς και άρθρα βασίζεται αυτή η δράση η οποία ελήφθη στα σύνορα. Δεύτερη και τελευταία μου ερώτηση είναι μας είπατε, μας λέτε ότι εμείς θα δούμε την Κροατία να εντάσσεται στον χώρο Σέγγεν. Νομίζω είναι πολύ καλά μαντάτα αυτά. Όμως διαρωτώ με ποια είναι η ανάλυση που κάνετε σε σχέση με τους μετανάστες ε, που μετακινούνται μέσω Δυτικών Βαλκανίων και μέσω Μακεδονίας ε, καθοδόν προς ε, τον χώρο Σέγγεν βλέπουμε ότι καταλήγουν στην Ουγγαρία και από εκεί προσπαθούν να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς την Ευρώπη και θα μπορούσαμε, εγώ θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα μπορούσε να υπάρξει κάποια μετάθεση όσον αφορά δρομολόγια. Αν τώρα η Κροατία θα μπορούσε να είναι το εφαλτήριο από πλευρά Σέγγεν. Εξαρτάται από, το, από πού κοιτάζει κανείς και προσεγγίζει το θέμα. Ποια είναι η ανάλυση σας αυτών των μεταναστευτικών ροών που θα, θα μπορούν να διοχετεύουν μέσω Κροατίας αν ενταχθεί στη Σέγγεν η Κροατία. Ευχαριστώ για το σημείο προς εμένα θα το θέσω προς τους συντονιστές, θα το εγγράψω, θα, βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη Επόμενο, η κυρία Μέερ παρακαλώ. Ε, ehm, Ευχαριστώ πρόεδρε. Ακούγοντας ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διαβάζοντας αυτή την έκθεση ένα συμπέρασμα μπορεί να διατυπώσει κανείς. Δεν λειτουργεί σωστά ο χώρος Σέγγεν για χιλιάδες μετανάστες. Η ασφάλεια των κρατών μελών απειλείται Υπάρχουν τεράστια προβλήματα στο Καλέ και στο Χουκ Φαν Χόλαντ με εκείνους που προσπαθούν ε, να περάσουν από τα κράτη-μέλη και να καταλήξουν ε, εκεί όπου επιθυμούν με μεθοριακούς συνοριακούς ελέγχους που δεν είναι πολύ αποτελεσματικοί και στην Σύνοδο ε, είναι λόγος για ε, εκατοντάδες χιλιάδες ε, συλλήψεις ε, για άλλους που μετέφεραν ναρκωτικά, για άλλους που δεν είχαν άδεια διαμονής. Δεν θα έπρεπε η όλη πολιτική να αναθεωρηθεί, να αναδιαρθωθεί και να αρχίσουμε να έχουμε συνοριακούς ελέγχους. Αν πράγματι δεν λειτουργεί το Σέγγεν, γιατί δεν το αναθεωρούμε και δεν το μεταρρυθμίζουμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε προλαλήσαντες αρκετοί ανέφεραν αυτό το θέμα που ήθελα εγώ να πω αλλά, να αναφέρω, αλλά σε σχέση με τα μέσα για τους ελέγχους στα σύνορα γίνονται κάποιοι έλεγχοι σε σχέση με την Αυστρία προς τα Ιταλικά σύνορα. Αυτό που γίνεται, αν συμβαίνει αυτό, εγώ πιστεύω ότι είναι απόλυτα κατανοητό βέβαια, αλλά θα ήθελα να μάθω ποια ακριβώ είναι η νομική βάση για να γίνεται αυτό και ποια είναι ακριβώς η φύση αυτών των ελέγχων στα σύνορα. Επίσης και μετά τη σύνταξη αυτής της έκθεσης Κάποια κράτη-μέλη ζήτησαν να πάψει να ισχύει ο μηχανισμός αυτός. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και η Σιλβή Γιώμ τελευταία παρακαλώ. Ευχαριστώ. Και εγώ αισθάνομαι ότι με αφορά αυτή η συζήτηση παρόλο που δεν έχω γράφει στο κατάλογο Δεν θέλω να παρέμβω στο έργο των γαλλικών αρχών, όμω για τα θέματα αυτά, τα θέματα Σέγγεν, που είναι ευαίσθητα γιατί αφορούν τα σύνορα. Έχουμε την εντύπωση ότι ο ένα πετάει την ευθύνη στον άλλον με του ανθρώπου να πηγαίνουν έρχονται μεταξύ των σύνορων. Και η προβολή από τα μέσα μαζική ενημέρωση δυστυχώ δυσκολεύει τα πράγματα. Θα συμφωνήσω όμω, είπε η Μαρία Κριστίν Βεριά, ακόμη και αν αυτό σα εκπλήσει. Ξέρουμε ακριβώ γιατί μιλάμε όταν μιλάμε για Σέγγεν. Δεν είμαι βέβαια Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Και βλέπω ότι και ο Κάρλος Κοέλιο συμφωνεί με αυτή την εντύπωση. Θα ήταν χρήσιμο πάντως η Επιτροπή να ε, κοιτάξει, να ερευνήσει τι γίνεται με τις γαλλικές αρχές και αν, υπάρχουν, υπάρχει παραβίαση των ευρωπαϊκών κανόνων. Διότι ποιος ε, αναφέρεται βεβαίω αυτέ τι δράσει, δεν θα πρέπει να ξεχνά και τι γαλλοϊταλικέ συμφωνίε για τα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών. Οι ξένοι που μπορεί να περνάνε τα σύνορα προ τη Γαλλία μπορεί με τη διαδικασία επανεισδοχή να επιστρέφουν. Αλλά θα πρέπει να δούμε αν υπάρχει παραβίαση. Σε αυτή τη φάση ε, έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχει παραβίαση από την πλευρά των γαλλικών αρχών, όμω γενικώ αυτή η κατάσταση δυστυχώ είναι πολύ δυσάρεστη και για τα άτομα και για τα κάτι μέλη που αφορά το φαινόμενο. Ευχαριστούμε και κύριο Δεκόιστερ για μια συντομότατη ε, τοποθέτηση. Ξέρω ότι έχετε πάρα πολύ λίγο χρόνο για να απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις, αλλά τέσσερα λεπτά το πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η σειρά ερωτήσεων που διατυπώθηκε θα απαντηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Για παράδειγμα, όσον αφορά τους αριθμούς των ποσών του προϋπολογισμού όσον αφορά το τρίτο, πρόγραμμα τρίτονας, τρίτων και ποσειδών. Θα δοθούν λοιπόν επακριβείς απαντήσεις όσον αφορά τα, τις προτάσεις για τον προϋπολογισμό όπως έχουν διατυπωθεί. Εντάχει κάποια άλλα σχόλια. Η έκθεση για τις δευτερογενείς κινήσεις ε, διατύπωσε ένα ερώτημα σχετικά ο κύριος Κοέλιο με αυτό θα είναι διαθέσιμα αυτά τα στοιχεία συντομότατα τις επόμενες εβδομάδες από την Frontex και την Europol και θα βρεθούν στη διάθεσή σας σαφώς. Επίσης το θέμα και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τις νέες ευθύνες που έχει δεν θα επισέθω σε λεπτομέρειες, αλλά πράγματι η ενίσχυση των στελεχών των αντίστοιχων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνέβη, έγινε ήδη. Είναι πολύ μεγάλο αυτό το έργο, πολλή δουλειά συνεπάγεται, αλλά οι πρώτες εμπειρίες, τα πρώτα βιώματα είναι θετικά. Έχουμε και το θέμα των πρόσφατων γεγονότων αν μου επιτρέπετε επ' αυτού πρόεδρε, δύο λόγια μόνο. Όλοι ακούσαμε δηλώσεις που έγιναν και τις επανέλαβε ο τύπος για κλείσιμο λέει συνόρων από την Γερμανία, Ελβετία, Αυστρία, Γαλλία. Καθότι γνωρίζουμε δεν υπάρχει κάποια, κάποιο τέτοιο κλείσιμο συνόρων με την εισαγωγή ελέγχων όσον αφορά τα εσωτερικά σύνορα στόχοθετημένα όσον αφορά τα μέλη της ε, ΛΥΜΠΕ στις ερωτήσεις που έγιναν. <clears throat> Δεν υπήρξε χρήση της ε, ρήτρας ασφαλείας Safeguard Clause. Δεν υπήρξε κάποια ειδοποίηση για επανεισαγωγή τέτοιων ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα. Και πρέπει να σας επιστήσω την προσοχή σας, δεν επιτρέπονται τέτοιοι έλεγχοι σύνοριακοί στα σύνορα αστυνομικοί έλεγχοι επιτρέπονται σε όλη την επικράτεια, ακόμα και σε περιοχές και περιφέρειες κοντά στα εσωτερικά σύνορα. Προφανώς πιθανότατα η διαφορά μεταξύ ελέγχων συνοριακών και άλλων αστυνομικών ελέγχων μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο για διδακτορική διατριβή οι διαφορές μεταξύ τους. Ωστόσο, το πλαίσιο αυτό επιτρέπει στα κράτη-μέλη να ασκούν αστυνομικούς ελέγχους και στο άρθρο 21 διατυπώνει μια σειρά όρων και προϋποθέσεων για να συμβεί κάτι τέτοιο. Όταν θα έχουμε ίσως περισσότερο χρόνο για μια σε μεγαλύτερο βάθος συζήτηση, αυτό θα μπορούσε σε μεγαλύτερο βάθος να συζητηθεί και να αναλυθεί μεταξύ μας. Εν πάση περιπτώσει, εχθέ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με βάση τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, είχε συναντήσει με υπουργού ε, των κρατών μελών, ώστε να γίνει μια διακρύβωση των στοιχείων, ποιου είδου ε, έλεγχοι, με ποια συχνότητα κτλ. γίνονται και μετά θα διατυπωθεί η θέση, η τοποθέτηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμω το κλείσιμο συνόρων σε σχέση με αυτά τα οποία αναφέρθηκαν δεν έγινε. Δεν έγινε τέτοιο κλείσιμο συνόρων. Σέγγεν αποτελεί μέρος του προβλήματος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι πρέπει να είναι μέρος της λύσης διότι έχει θεσπιστεί μια ολόκληρη σειρά όρων για συνεργασία, για κοινέ προδιαγραφές και διατάξεις που πρέπει να εφαρμόζονται από όλα τα κράτη-μέλη και αυτό θα διευρύνει την ασφάλεια αν γίνει σωστά. Επιτρέψτε μου ρητορικά να θέσω το ερώτημα, απαντώντα σε κάποια ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα του Σέγγεν. Πραγματικά πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση <clears throat> δεν θα υφίστατο μεταναστευτικές ροές αν υπήρχαν έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα. Okay, thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Όπως είπα συνάδελφοι, θα μπορούσαμε να είχαμε μια συζήτηση πολύ πιο σε βάθος και πολύ πιο ε, μεγάλη, όμως δεν έχουμε χρόνο. Σας ευχαριστώ λοιπόν που είστε πειθαρχημένοι. Σίγουρα τα ζητήματα για το Σέγγεν θα ανακύψουν και στις 10.45 που θα έχουμε τη Λετωνική Προεδρία. Ας πάμε στο σημείο 13. Ίση μεταχείριση των ανθρώπων ανεξαρτήτως του σεξουαλικού τους προσανατολισμού, του φίλου, της θρησκείας τους, ε, της ηλικία και το καθεξής. Ε, θα ακούσουμε την κυρία Σολβίτα Βεβέρε, η οποία είναι διευθύντρια της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο για την πρόταση οδηγίες για την ήσυχη μεταχείριση ανθρώπων ανεξαρτήτως ε, φύλου κλπ. Ε, η συγγήτρια για... στην Επιτροπή μας είναι η κυρία Λούνατσεκ. Η οδηγία αυτή αποκαλείται οριζόντια οδηγία. Κυρία Βεβέρε, είστε εδώ, είστε έτοιμοι. Δεν θα κάνω άλλες εισαγωγικές παρατηρήσεις για να έχετε περισσότερο χρόνο. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Κυρία Λούνατσεκ, κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη που ενδιαφέρεστε για αυτό το φάκελο. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που βρίσκομαι στην Επιτροπή σας σήμερα. Και χαίρομαι διότι έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το σημαντικό ζήτημα της ίσης μεταχείρισης. Η πρόταση της Κομισιόν για μια νέα οριζόντια οδηγία στο το πεδίο αυτό συζητείται στο Συμβούλιο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είχα την ε, δυνατότητα να συμμετάσχω στο Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ του Δεκεμβρίου και λόγω του αδιεξόδου στο Συμβούλιο, του τόσο μακρού αδιεξόδου, θεωρεί η Ιταλική Προεδρία, θεώρησε ότι πρέπει να έχουμε ενισχυμένη συνεργασία, να εξερευνήσουμε όλες τις άλλες εναλλακτικέ. Κατά τη διάρκεια της υπουργική συζήτησης κατέστη σαφές ότι παραμένει ισχυρή η στήριξη του Συμβουλίου για ποιο πράγμα, για το να συνεχιστεί η δουλειά για την πρόταση. Η ίση μεταχείριση ήταν ένας από τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό ορίζεται στις συνθήκες. Συνεπώς υπήρχε έλλειψη στήριξης να ακολουθηθεί η οδός της ενισχυμένης συνεργασίας. Ωστόσο, η συζήτηση κατάφερε να διεγείρει τελικά τις διαπραγματεύσεις και να τις ε, πυροδοτήσει. Όμως, όπως ε, καταλαβαίνετε, είναι περίπλοκο το ζήτημα και γι' αυτό χρειάζονται περαιτέρω συζητήσεις και διευκρινήσεις για να επιτευχθεί απαραίτητη ομοφωνία οι προεδρίες το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να ακολουθούν τις απόψεις όλων των κρατών μελών, ακόμα και των κρατών μελών που ευρίσκονται σε θέση ε, μειοψηφία. Όμως, κατά τη διάρκεια της εξάμενης Λετωνικής Προεδρίας κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να προχωρήσουμε στο φάκελο αυτό. Και θα ήθελα να σας κάνω μια επισκόπηση της δουλειάς που έγινε στην ομάδα εργασίας το Φεβρουάριο και το, από το Φεβρουάριο μέχρι το Μάιο. Η Λετωνική Προεδρία υπέβαλε φρέσκες προτάσεις διατύπωσης ε, οι οποίες ασχολήθηκαν κυρίως με το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Η διαίρεση των αρμοδιοτήτων μεταξύ κρατών μελών και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είναι για κάθε θέμα το πιο κρίσιμο σημείο και πάντοτε πρέπει να βρούμε σωστές διατυπώσεις όσον αφορά στην κοινωνική προστασία μεταξύ άλλων. Και δουλέψαμε και πάνω στην έννοια της διάκρισης και πιο συγκεκριμένα ε, ασχοληθήκαμε με τη μεροληψία λόγω της ηλικία και προσπαθήσαμε να έχουμε ισορροπία μεταξύ από τη μία της προστασίας κατά των διακρίσεων, αυτό εδρεώνεται με την οδηγία και από την άλλη πλευρά ε, με τα μέτρα που ε, υπάρχουν στην εθνική νομοθεσία. Επιπροσθέτως, η Λετωνική Προεδρία κυκλοφόρησε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο απευθύνει σε όλες τις αντιπροσωπίες καλώντας τις να διευκρινίσουν τις θέσεις τους και όσον αφορά στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και όσον αφορά στο ποιο πιστεύει κάθε αντιπροσωπεία ότι είναι το πιο σημαντικό ε, εκρεμές ζήτημα και ως προς το ε, ποιο είναι το επιθυμητό χρονοδιάγραμμα για κάθε αντιπροσωπεία. Γιατί το κάναμε αυτό και μοιράσαμε το ρηματολόγιο για να δώσουμε συνέχεια στη δουλειά που έχει ήδη γίνει και για να πλησιάσουμε ακόμα περισσότερο την απαιτούμενη ομοφωνία. Συγκεντρώσαμε τις απαντήσεις, τις βάλαμε σε ένα ενιαίο έγγραφο το οποίο θα είναι χρήσιμο υπόβαθρο για την επόμενη Προεδρία επάνω στο φάκελο αυτό. Τώρα, η Λετωνική Προεδρία υπέβαλε μια έκθεση προόδου στο Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ, το οποίο συνέρχεται αύριο στις 18 Ιουνίου στο Λουξεμβούργο. Και συμπερασματικά θα ήθελα να, αντιμετω... να σας μιλήσω για τους περιορισμούς της Λετωνικής Προεδρίας και της κάθε Προεδρίας. Από... Όταν απαιτείται ομοφωνία ε, σε ένα θέμα δεν μπορούμε να προσαρμόσουμε την υφιστάμενη νομοθεσία μέχρι ότου συμφωνήσουν όλα τα κράτη-μέλη. Και ε, οι προτάσεις έχουν ληφθεί από το 2008 που είναι ανοιχτός αυτός ο φάκελος και ελπίζω ε, κάποια στιγμή να επιτευχθεί συμφωνία. Thank you very much. This is, um, again... Ευχαριστούμε πολύ. Συνάδελφοι, όπως αναφέρθηκε, πολλοί από μας έχουν δουλέψει στην οδηγία αυτή, γιατί ήδη συζητιέται από το 2008. <coughs> Θα δώσω πρώτα το λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Λούνατσεκ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τη Λετωνική Προεδρία που προσπάθησε να προχωρήσει και να έχει αυτή τη διαβούλευση με τα κράτη-μέλη και με αυτή την έκθεση πρόοδου που μας διέθεσε και ελπίζω ότι αυτό θα είναι η βάση με την οποία θα προχωρήσουμε μελλοντικά καθότι κατανοώ και δεν θέλω να επισέθω σε όλες τις λεπτομέρειες όσων έχουμε τώρα στη διάθεσή μας αλλά από ό,τι κατανοώ υπάρχει μεγάλη ανησυχία στα κράτη-μέλη όσον αφορά τα θέματα επικουρικότητας και όπως είπατε για τα θέματα κοινωνικής προστασίας και θέματα παιδείας εκπαίδευσης. Και κατανόησε επίση ότι έχουν κάποια προβλήματα με την, ε, το θέμα της νομικής βεβαιότητας και ασφάλειας κάποια κράτη-μέλη. Όμως ε, ελπίζω ότι αυτό δεν θα έπρεπε να είναι το κύριο πρόβλημα. Κανόνας λόγο για τα, τις ανησυχίες για την επικουρικότητα με εκπροσώπους ε, των κρατών μελών με τους οποίους έχω συζητήσει πολύ καλό είναι να τα αναφέρουμε όλα αυτά και να συγκρίνουμε τι συμβαίνει με την οδηγία για την απασχόληση και την ε, φιλετική ισότητα. Συμμετέχοντας σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις από τα κράτη-μέλη δεν υπήρξαν κάποιες ανησυχίες όσον αφορά το θέμα της επικουρικότητας. Και τώρα είναι παρόμοιο αυτό. Παρόμοιο, μόνο, η κατάσταση παρόμοια μόνο για διαφορετικές ομάδες ε, ατόμων. Και όταν κάνουμε λόγο για την οδηγία αυτή, ελπίζω ότι αυτές οι ανησυχίες ε, δεν θα διαπιστωθεί ότι έχουν λόγο ε, να υφίστανται περαιτέρω. Κάνοντας λόγο για την παιδεία και την εκπαίδευση γνωρίζουμε ότι είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών βεβαίως αυτό το θέμα. Όμως σε σχέση με τις ανησυχίες ότι λένε κάποιοι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να επιβάλλει το πόσο και με ποιο περιεχόμενο θα συντάσσονται ε, τα διάφορα εγχειρίδια, βιβλία ε, των σχολείων. Θέλω να αναφέρω τι σημαίνει η μη εφαρμογή αυτής της οδηγίας με κάποια παραδείγματα. Σε σχέση με κάποιο ε, παιδί που θέλει να πάει στα γενέθλια του ενός κοριτσιού και που θεωρείται ότι ε, αυτό το παιδί μπορεί να, θεω... Ε, να αντιμετωπίζεται ως ομοφιλόφιλος. Ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν εδώ επιπτώσεις όσον αφορά παράδειγμα ένας πατέρας ο οποίος εργάζεται μόνο με εργασία μερικού χρόνου και δεν υπάρχει κανένας τρόπος από πλευρά σχολείου να ε, συζητηθούν αυτά τα θέματα ε, σεξουαλικού προσανατολισμού και επιλογών για παράδειγμα. Τότε στην παιδεία και εκπαίδευση φυσικά πρέπει να υπάρχουν στοιχεία που να πληροφορούν τα παιδιά για το τι ε, συνεπάγεται και περί πρόκειται το θέμα των σεξουαλικών προσανατολισμών σε σχέση με τα αγόρια και τα κορίτσια που διαφορετικά δεν θα υφίστατο. Να δώσω και ένα παράδειγμα σε σχέση με την προσπελασιμότητα σε δημόσιους χώρους. Στη δική μου χώρα, την Αυστρία, πρόσφατα τον Ιανουάριο, ένα ζεύγος λεσβίων ήθελε να πάει σε ένα από τα παραδοσιακά καφενεία της ε, Βιέννης και όταν συναντήθηκαν φιλήθηκαν και αποφάσισε ο ιδιοκτήτης ή η ιδιοκτήτρια του καφενείου ότι δεν έπρεπε να γίνεται αυτό, δεν ήταν ηθικό και τις έδιωξε από εκεί. Τώρα, αν αυτό είχε συνέβαινε <coughs> για παράδειγμα ένα ε, ζευγάρι ε, ε, μαύρων είχαν φιληθεί και είχαν εκδιωχθεί θα μπορούσαν να προσφύγουν στα δικαστήρια και να πούν ότι αυτό αποτελεί αρνητική διακριτική μεταχείριση. Αυτό δεν μπορούσαν να το κάνουν οι λεσβίες το ζευγάρι αυτό. Αυτό πάλι αποτελεί ένα παράδειγμα το ότι τα κράτη-μέλη πρέπει πραγματικά να εφαρμόζουν τα θέματα μη αρνητική διακριτική μεταχείρισης. Όμω δεν πρόκειται εδώ για θέμα επικουρικότητα αλλά για θέμα ισότητα. Είναι πάλι επίση πτήθεται το θέμα του κόστου το παράδειγμα της Ιρλανδίας που δείχνει ότι έγινε μία μελέτη μετά από το νομοθέτημα, μετά από 12 χρόνια που ίσχυε η νομοθεσία για την ίση μεταχείριση. Και όλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχει ένα κόστος, αλλά η σύγκριση για την διεύρυνση της προσπελασιμότητας για άτομα με ειδικέ ανάγκες ε, <clears throat> αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να θεωρηθεί ως πρόσκομα ή ε, σημαντικό εμπόδιο. Τώρα, σε σχέση με τα όσα αναφέρονται το Δεκέμβριο για το ότι απορρίφθηκε η διευρυμένη συνεργασία από τα κράτη-μέλη, το εκτιμώ, την αναφορά. Η ισότητα η οποία κατοχυρώνεται στις συνθήκες και στην χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν μπορούμε επιλεκτικά να επιλέξουμε κάποια θέματα και να λέμε για αυτά μπορεί να ισχύει η ισότητα για άλλα όχι. Λοιπόν, ίσως τώρα όμως μια ερώτηση προς εμάς και εδώ στην Ευρωβουλή έχουμε ευρύτατη συνένεση για αυτή την οδηγία. Τι γίνεται λοιπόν με το να ζητούσαμε από το Συμβούλιο επίσης να προσκαλέσει ευρωβουλευτές και ευρωβουλευτίνες να διεξαχθεί μια συζήτηση με αυτούς και να τύχει συνέχεια το θέμα των ανησυχιών και μελημάτων τους διότι θα μπορούσαν να αρθούν αυτές, ε, αυτά τα προβλήματα και ανησυχίες αν υπήρχε άμεση επαφή θα το εκτιμούσαμε αν γινόταν αυτό από την Προεδρία. Δεν είναι ανάγκη να γίνεται αυτό υπό τον τύπο και μορφή των συναντήσεων, των συνεδρίων, συνεδριάσεων του Συμβουλίου. Θα μπορούσε να εξευρεθεί και μια άλλη ε, μορφή, ένα άλλο είδο επαφών, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα και να αρθούν αυτέ οι ανησυχίε των Ευρωβουλευτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ουρίκε. η κυρία Κοράτσα Μπιτ, Γιώμ, Κερκόπ, Υπάρχει κάποια κούραση μετά από όλη αυτή, όλο αυτό το γύρο. Εντάξει η Χέργα, ο κύριος Στίβενς, εντάξει. Okay, that's the list. Um, can I just close the list because I don't want to... Uh... Αυτός ήταν ο κατάλογος, να τον κλείσω διότι θα ήθελα να περάσουμε στα συμπεράσματα της Προεδρίας που όλοι αναμένουμε διακαώς. Να ξεκινήσουμε με την κυρία Κοράτσα Μπιλτ. Κυρία Κοράτσα, μία ερώτηση. αν δεν σας πειράζει και αν με ακούει το Συμβούλιο, να κάνω ακόμα τη δική μου ερώτηση. Τέλος πάντων, ε, δεν είναι πολύ σημαντικό ίσως τη Δευτέρα, ούλη ε, συζητήθηκε το θέμα του πεδίου και της πλατφόρμας και κάπως διευρύνθηκε και σε συζήτηση με το Συμβούλιο της Ευρώπης και άλλους συναδέλφους. Υπήρξε όμως δυσαρέσκεια, κάποια σχετική δυσφορία για το θέμα του κόστους. Είπατε ότι πρέπει να υπάρχει μια δικημενική προσέγγιση σε όλες τις χώρες που εκπροσωπούνται εδώ Θα ήθελα την δική σας την ε, τοποθέτηση γι' αυτό. Υπάρχουν αρκετά στοιχεία. Το έχετε μελετήσει. Θα θέλαμε τη δική σας πρόπτικη εφόσον βρισκόμαστε στο τέλος προεδρίας. Δεν μπορείτε βεβαίως να αναλάβετε πλήρως την ευθύνη αλλά η άποψη των τόσο αντιπροσωπευτικών οργανισμών που συναντήσαμε τη Δευτέρα εδώ για το θέμα αυτό στις Βρυξέλλες ήταν αυτή. Η κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα συμφωνήσω με τα σχόλια της συγκεκριάς της κυρίας Λούνατσεκ και θα συμφωνήσω με την δυσαρέσκεια για την διαδικασία αυτή που τόσο πολύ έχει απομονωθεί. Την τελευταία φορά που το συζητήσαμε ήταν τον Νοέμβριο Καλωσορίζω όλε τι προσπάθειε που έχει καταβάλει η Λεπτονική Προεδρία. Σα ευχαριστούμε πολύ πραγματικά. Θα, θα ήταν ωραία να δούμε και χειροπιαστά αποτελέσματα από το ερωτηματολόγιο. Διότι είναι σημαντικό για λόγου διαφάνεια. Για να δούμε ποια είναι τα προβλήματα, ποιε οι ανησυχίε στο Συμβούλιο για την επικουρικότητα και για αυτό που πολύ σωστά περιέγραψε η Ουρίκε. Γιατί να μην είναι θέμα η επικουρικότητα. Μιλούμε για μια μεγάλη αρχή μη διακριτική μεταχείριση που θα πρέπει να περνά όλη την εθνική νομοθεσία. Είναι οδηγία, δεν είναι κανονισμός. Η επικουρικότητα δεν είναι επιχείρημα. Και το θέμα του κόστους, εντάξει, υπάρχουν σοβαρές ε, ανησυχίες, το καταλαβαίνω, ιδίως για τον ιδιωτικό τομέα, όμως δεν είναι η στιγμή στην Ευρώπη να περάσουμε σε μια κοινωνία που να συμμετέχουν όλοι με τον ίδιο τρόπο. το ποιε είναι οι συγκεκριμένε ανησυχίε μα. Είναι θέμα χρόνου. Τουλάχιστον το Συμβούλιο εγκατέλειψε την ιδέα της ενισχυμένης συνεργασίας. Όμως και πάλι δεν φτάνει αυτό. Να πω ότι είναι πολύ σημαντικό σε αυτή τη φάση όπου έχουμε τοποθετήσεις με λόγια μίσους, ε, με πολιτικούς που καταδικάζουν συγκεκριμένες ομάδες προσώπων, με εξτρεμιστικές τάσεις στην Ευρώπη. Η οδηγία αυτή για την ίδια κριτική μεταχείριση γίνεται όλο και πιο επίκαιρη. Ακούσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σχολιάζει και προηγουμένω τη διαφορά μεταξύ ελέγχου των συνόρων και ε, παρουσίαση των αστυνομικών στα σύνορα. Όμω, τι γίνεται με την ε, καταγραφή των θρησκευτικών πεπιθήσεων κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ελέγχων. Αυτό και από τη σκοπιά τη μετανάστευση είναι ένα πραγματικό πρόβλημα. Μπορεί να υπάρξει διακριτική μεταχείριση και βάση τη θρησκεία και των πεπιθήσεων. Και η τελευταία μου παρατήρηση είναι ότι πραγματικά ελπίζω κάποια από τα κράτη-μέλη να μην χρησιμοποιούν την επικουρικότητα ή το κόστος ως δικαιολογία για να ε, μην παραχωρήσουν ίσα δικαιώματα στους ε, ΛΟΑΔ. Ευχαριστούμε κυρία Γκουγιόμ. Ευχαριστώ και εγώ θα εκφράσω τη δυσαρέσκειά μου όπως οι συνάδελφοι. Η δυσφορία είναι και δική μας για το κείμενο αυτό που δεν σταματά να γνωρίζει εμπόδια. Όμως βλέπουμε ότι η διακριτική μεταχειρήση όχι απλώς δεν αναχαιτίζεται στην Ευρώπη, όλο και πιο πολύ μας ε, κάνει να βλέπουμε ότι πρέπει να κρούσουμε τον κόρονα του κινδύνου. Είναι λοιπόν ανάγκη να προασπίσουμε τις ευρωπαϊκές αξίες για την εικόνα και το καλό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν συμμερίζομαι πολύ την ιδέα της Ούρλικε για την ενισχυμένη συνεργασία λέγοντας ότι είναι μια κακή λύση. Δεν ξέρω. Ήταν και ένα μέσο δράσης από το τίποτα, παρόλο που εγκαταλείφθηκε ως ιδέα. Εάν δεν γίνει τίποτα, πού θα πάμε. Αρκεί να προσκαλούμε βουλευτές να συζητούν με το Συμβούλιο, δεν είμαι βέβαια. Ίσως λοιπόν θα πρέπει να πάρουμε θέση και για το τι συγκεκριμένη ε, κατάληξη θέλουμε να έχουμε. Θέλουμε να έχω η συζήτηση αυτών των θεμάτων. Ευχαριστούμε κύριος Κέπλε. Κύριε Πρόεδρε, βεβαίω καλωσορίζω αυτές τις εξελίξεις. Η ανάγκη για ισότητα και μη διάκριση είναι επιτακτική σε όλους τους τομείς στους οποίους αναφερθήκατε. Δεν μιλούμε μόνο για το σεξουαλικό προσανατολισμό, τις σεξουαλικές προτιμήσεις, μιλούμε για τις αναπηρίες, για τις διακρίσεις που πλήττουν με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους το σύνολο της κοινωνίας. Πολλοί νέοι θεωρούν ότι ορισμένες φορές πρέπει να μεριμνούμε ιδιαίτερως για την κοινωνική πολιτική και ότι είναι τα κράτη-μέλη που έχουν αυτή την αρμοδιότητα. Εγώ θεωρώ ότι Κάθε φορά που γίνεται προσπάθεια να εφαρμοστεί μια τέτοια νομοθεσία, δεν αρκεί ως προσπάθεια. Οι νομοθέτες τείνουν να πιστεύουν ότι άπαξ και νομοθετήσουν έχουν κάνει τη δουλειά τους και δεν υπάρχει καμιά άλλη ευθύνη για τα ζητήματα αυτά και μπορούμε με, με φιλαρέσκεια να είμαστε ικανοποιημένοι για την πράξη μας. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Οι προκαταλήψεις και οι διακρίσεις παραμένουν ριζωμένες για πολλά χρόνια και δεν τελειώνει η δουλειά μας με την ψήφιση της οποιασδήποτε νομοθεσίας. Έχω ωστόσο ένα ερώτημα. Ε, μετά από τη συμφωνία, ποιες προοδοί αναμένονται στο εκπαιδευτικό κομμάτι, για την εκπαίδευση των ανθρώπων στην Ευρώπη και για τις διαδικασίες παράβασης, επί παραβάση. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος, χρειάζεται δράση στη βάση της κοινωνικής πυραμίδας για να καταπολεμήσουμε την ανισότητα και να προωθήσουμε την ανοχή, την ε, ανοχή στο διαφορετικό και την αποδοχή. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Ναι. Δεν υπάρχει εξέλιξη από το 2008 για τα θέματα αυτά. Προφανώ θα θέλαμε να δούμε κάποια χειροπιαστή δράση και μετά θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την πραγματική υλοποίηση. Η κυρία Ινφελτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι η τρίτη μου θητεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι η τρίτη θητεία κατά την οποία συζητούμε αυτό το φάκελο. Πόσε φορέ πρέπει να επανεκλεγώ για να δούμε αυτό το φάκελο να φτάνει ε, σε ένα ε, αίσιο τέλος. Ο πρόεδρος είναι η καλή στρατηγική σου Σοφία πάντως. Η Σοφία Ιντβελτ. Ας έχουμε μια ειλικρινή συζήτηση. Γιατί έχει κολλήσει αυτός ο φάκελος τόσα χρόνια. Όχι γιατί υπάρχουν τεχνικά εμπόδια. Με τα ίσα δικαιώματα για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά έχει κολλήσει ο φάκελος γιατί τα κράτη-μέλη δεν το επιθυμούν. Αν ήθελαν την ίση μεταχείριση θα την έκαναν σήμερα ακόμα και χωρίς την οδηγία. Επομένως, το βασικό πρόβλημα εδώ είναι η έλλειψη πολιτικής βούλησης ορισμένα κρατημέλη. Το αποκαλούν επικορικότητα, αλλά αυτό που λένε είναι ότι θέλουμε την ελευθερία εμείς να διακρίνουμε όποιο νομίζουμε. Ας το συζητήσουμε αυτό και απευθύνομαι σε όλες τις πολιτικές ομάδες, γιατί όλες οι πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θέλουν την ίση μεταχείριση. Δεν είναι και τόσο δύσκολο, δεν είναι πυρηνική επιστήμη. Ορισμένα κράτη-μέλη δεν θέλουν στα αλήθεια την ίση μεταχείριση. Γίνεται λόγος για παράδειγμα για το κόστος των ίσων δικαιωμάτων. Π.χ όταν ε, μιλούμε για τη διάκριση με βάση την αναπηρία ή την ηλικία. Έχουμε αυτή την ε, έκθεση τόσο πυκνή και πολυσέλιδη. Ε, λοιπόν, έχουμε υπολογίσει το κόστος της διάκρισης της ανισότητας. Δηλαδή να μην υπολογίσουμε μόνο το κόστος της ισότητας όταν εφαρμόζεται. Εγώ θέλω και έκθεση που να υπολογίσουμε το κόστος της ανισότητας όταν αυτή εφαρμόζεται. Από εκεί και πέρα να πω ότι ορισμένοι πολίτες θα είχαν δικαίωμα σε ίση μεταχείριση και άλλοι όχι δυστυχώς. Και τα κράτη-μέλη τελικά δεν λένε το οριστικό όχι, γιατί ξέρουν ότι αυτό θα αντίκητο στις συνθήκες. Και γι' αυτό τελματώνεται όλη αυτή η ιστορία με αυτό το φάκελο. Γνωρίζουμε ότι στην εκπαίδευση και στην υγεία είναι οι τομεί με τα μεγαλύτερα προβλήματα, κυρίως στην εκπαίδευση. Εκεί έχουμε διακρίσεις κάθε είδου και εμπόδια. Άλλωστε ακούστηκε και αυτό το περίεργο παράδειγμα όπου όπου ε, μαζικά υπήρξε ψηφοφορία υπέρ των γάμων ατόμων ιδίου φύλου και κάποιος ε, ε, ιερέας κάποιες εκκλησίες είπε ότι αυτό είναι τραγικό γιατί οι ψηφοφόροι σε μεγάλο βαθμό είχαν μορφωθεί σε καθολικά σχολεία. Ή άλλοι λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται να μας επιβάλλει την ισότητα. Αλλά εγώ απαντώ, η ισότητα είναι στις συνθήκες και κάθε χώρα προσχώρησε στη συνθήκη εθελοντικά. Ήθελε και ήρθε, ήθελε και μπήκε. Εν πάση περιπτώσει η δέσμευση για την ισότητα δυνατότητα πρέπει να είναι αταλάντευτη. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Παρακαλώ να είστε σύντομοι. Μάλλον παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη για τα περισσότερα προαναφέρθηκαν ήδη. Θα ήταν ενδιαφέρον να βλέπαμε αυτό το ερωτηματολόγιο για εμάς τους Ευρωβουλευτές να δούμε ποια προβλήματα και ανησυχίες υπάρχουν και ποια προσκόμματα. Επίσης θέλω να υποστηρίξω αυτό το οποίο προαναφέρθηκε. Σε μια κατάσταση όπως τη σημερινή τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα υπάρξει ένας χώρος ε, για τα κονδύλια, ε, για τη χρήση Frontex. Ε, τι θα κάνουμε με τους μετανάστες. Θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε επί θεμάτων για την ισότητα, για το συμφέρον των πολιτών μας. Θα ήθελα να υπάρξει αυτή η απάντηση, ότι δηλαδή εργαζόμαστε προς το, με στόχο την ισότητα για τα δικαιώματα του ανθρώπου και την ισότητα δεν κάνει τίποτα η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Και όπως προναφέρθηκε από προλαλήσαντες, Χρειαζόμαστε αυτή την οδηγία. Χρειαζόμαστε την ισότητα και την ίση Δεν την έχουμε ούτε στα σχολεία, ούτε στην καθημερινή δημόσια ζωή και υπάρχουν ομάδες που δεν προστατεύονται πλέον από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και χρειάζονται αυτή την νομοθεσία για να προστατεύονται και συμφωνώ με την κυρία Ιντφέλτ και εγώ θα ήθελα να ξέρω ποιο είναι το κόστος της μη ισότητας στην Ευρώπη είναι πολύ υψηλότερο από το κόστος της ισότητας σας ευχαριστούμε πολύ η παρακαλώ έχετε τον λόγο Σας ευχαριστώ πρόεδρε Ευχαριστώ Πρόεδρε. Με μεγάλη χαρά ακούσα από την Λετωνική Προεδρία το ότι <clears throat> δεν επελεγεί διευρυμένη συνεργασία και σε σχέση με την ομοφωνία πολύ καλά πότε θα επιτευχθεί αυτή η ομοφωνία γιατί επί 8 χρόνια διαρκεί όλη αυτή η διεργασία και δεν έχει ολοκληρωθεί το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποια συμφωνία για το θέμα της αρχής της ισότητας είναι κοιλίδα, μελανώνει την, ε, ε τις επιδόσεις ε, του Συμβουλίου. Όλοι πρέπει να την χάνουν ίση μεταχείρισης. Πρέπει να ληφθεί επιτέλους μια απόφαση. Γνωρίζω ότι πρόκειται για ένα τεχνικού χαρακτήρα ζήτημα, αλλά η αρχή ότι όλοι είναι ίσοι είναι μια θεμελιώδης βασική αρχή της Ευρώπης. Αν λοιπόν αυτό το δεχόμαστε παρακαλώ να κάνουμε κάτι, να κάνετε κάτι το δυνατόν ταχύτερα. Επίσης ενδιαφέρομαι και για κάτι άλλο για τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου. Σε σχέση με το ερωτηματολόγιο, θα ήθελα να τα δω σε σχέση με αυτό το ερωτηματολόγιο και να δω ποια κράτη-μέλη δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους εδώ. Και έγινε και λόγος για το θέμα του κόστους. Κάποιες χώρες φοβούνται ότι θα υπάρχουν κόστη αν υπάρξει λέει μια οδηγία για την ίση μεταχείριση. Και όπως άλλοι συνάδελφοι ανέφεραν, το να αποκλείουμε ανθρώπους κοστίζει τεράστια ποσά. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το κόστος του αποκλεισμού. Εντάξει, κάνουμε λόγο για 10% του πληθυσμού μας εδώ συνολικά. Εκεί φίλοι, συγγενείς ε, υφίστανται όλες αυτές τις επιπτώσεις. Θα πρέπει λοιπόν πραγματικά να δούμε ότι ακόμα και ένα τέταρτο του πληθυσμού αποκλείονται συνολικά. Δεν μπορούν ούτε στον κινηματογράφο να πάνε, ούτε στο εστιατόριο όλοι μαζί. Δεν μπορούν να μπουν σε ένα λεωφορείο, σε ένα τρένο. Δεν μπορούν να κάνουν ένα τηλεφώνημα να κάνουν κάποιο άθλημα. Είναι οικονομικές απώλειες όλα αυτά και πρέπει να υπολογιστεί το κόστος αυτών των οικονομικών απώλειών. Και θέλω να υποστηρίξω το αίτημα να υπολογίσουμε το κόστος της μη ίσης μεταχείρισης. Όταν θα το έχουμε διαπιστώσει τότε θα μπορούμε να πάμε παραπέρα. Υπάρχουν μελέτες, ναι, αλλά πότε θα υπάρξει επιτέλους αυτή η οδηγία που πρέπει να εγκριθεί. Σε ευχαριστούμε. Είναι μια εξαιρετική συνεισφορά και ένα εξαιρετικό σημείο αφετηρίας. Λοιπόν, και για τους συναδέρφους ε, που σε σχέση με τα θέματα της Προεδρίας θα ήθελα να περάσουμε αμέσως στην Επιτροπή αν μπορείτε να είσαστε σύντομοι λυπούμε που σας πιέζω να είσαστε σύντομοι για αυτό το σημαντικό θέμα αλλά έχετε τον λόγο παρακαλώ Σας ευχαριστώ θα είμαι πολύ σύντομος απλώς να υπογραμμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, παραμένει αφοσιωμένη στην πρόθεση αυτής της πρότασης όπως και στο παρελθόν Έχουμε διαφορετικά κομματάκια για την ίδια κριτική μεταχείριση και την ισότητα στο ίδιο παζλ. Αυτό είναι το κομματάκι που λείπει για να ολοκληρωθεί η προστασία μα κατά τη διακριτική μεταχείριση ε, στον χώρο εργασία και παντού όπω προβλέπει το 19 τη συνθήκη. Γι' αυτό και ο πρόεδρο Γιούγκερ το προέλεπε στι κατευθυντήριε γραμμέ για την εντολή αυτή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το θεώρησε, το χαρακτήρισε απόλυτη προτεραιότητα προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες και να πείσουμε τα διστακτικά κρατημέλη να αφήσουν τις αντιστάσεις του. Ε, και θα φροντίσουμε να έχουμε τι απαραίτητε διμερεί επαφέ ε, στο επίπεδο των κρατών μελών, μεταξύ των επιτρόπων και των υπουργών των ενδιαφερομένων κρατών μελών, διμερεί επαφέ με τα κράτη-μέλη που δυσκολεύονται. Νομίζω ότι και οι πολιτικές προτεραιότητες και ε, οι δυσκολίες, οι τεχνικές δυσκολίες κάποιων κατών μελών μπορούν να αντιμετωπιστούν. Ε, θα έχουμε λοιπόν συνομιλίες και σε στενή συνεργασία με τις προεδρίες ε, εντός των οποίων και η λαπτονική προκειμένου να προωθήσουμε αυτό το θέμα. Το Συμβούλιο Κοινωνικών Υποθέσεων του περασμένου Δεκεμβρίου εκφράστηκε πολιτική βούληση το θέμα αυτό να προωθηθεί και η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών μελών έχει τη διάθεση η οδηγία αυτή να εγκριθεί. Μιλάμε για ένα πολύ μικρό αριθμό κρατών μελών που διαφωνούν και προσπαθούμε να τους μεταπίσουμε. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για την κοινωνική προστασία και την ε, εκπαίδευση. Έχουμε κάνει πολλά σε συνεργασία με τη Λετωνική Προεδρία για το χώρο της ε, προστασίας αυτής. Αλλά δεν έχουμε ακόμα τη συμφωνία των 28 κρατών. Δεν μπορούμε να το ανακοινώσουμε επισήμω. Είμαστε σχεδόν στου 28 και έχουμε δει χειροπιαστά αποτελέσματα επί Λετωνική Προεδρία. Για αυτό λοιπόν το πολύ δύσκολο θέμα, η μόνη μα επιλογή, εάν δεν θέλουμε να φτάσουμε σε απελπισία, είναι να εκμεταλλευτούμε κάθε δυνατότητα να προχωρήσουμε και αυτό το έχουμε καταφέρει με τη Λετωνική Προεδρία. Θα το κάνουμε και με την ερχόμενη Λουξεμβουργιανή. Και θα ακολουθήσουμε τι προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπω έχουν εκφραστεί. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ και την κυρία Βεβέρ. Ε, με συγχωρείτε που σα πιέζω. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα να απαντήσω στι ερωτήσει. Καταρχάς, να ευχαριστήσω για τα πολύτιμα σχόλια και συστάσεις. Είναι πολύ σημαντικό όλοι να συνδυάσουμε το έργο μας για να υπάρξει ομοφωνία και να γίνει δεκτή η οδηγία όπως ανέφεραν οι περισσότερες από τις αντιπροσωπείες. Πρέπει να προχωρήσει ως το δυνατόν γρηγορότερα. Ε, σε ό,τι αφορά τα σχόλια και τις ερωτήσεις που θα μεταβεβαστούν και στην επερχόμενη Προεδρία, να απαντήσω πρώτα απ' όλα στην ερώτηση για την γύρανση. αναφέρθηκαν ε, εξαιρέσεις ε, ώστε να μην χρησιμοποιείται η ηλικία ως ε, επιχείρημα επιβολή διαφορετικών τελών για τους πελάτες ή καταναλωτές. Εδώ η ερμηνεία διορθώθηκε γιατί ήταν ιδιαίτερα ευρεία. Επίσης για την κοινωνική προστασία και την εκπαίδευση η Προεδρία σκοπό έχει να ορίσει το πεδίο έτσι ώστε να είναι σαφές για τα κράτη-μέλη ποιες είναι οι αρμοδότητές τους για την χρηματοδότηση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και των εκπαιδευτικών συστημάτων. Θα συμφωνήσω με αυτό που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε εργαστεί αποτελεσματικά και αποτελεσματική δουλειά έχει γίνει στις περισσότερες αντιπροσώπειες. Οπότε έχουν γίνει βήματα πρόοδου προς την ομοφωνία. Και για τις σύντομε απαντήσεις του ερωτηματολογίου. Τα εκκρεμή ζητήματα. Σε αυτά να σταθώ. Συμφωνώ με την κυρία Λούνατσεκ ότι όλα τα εκκρεμή ζητήματα δεν έχουν καλυφθεί. Όμως, να σας επισημάνω και αυτό θα απασχολήσει και την ε, επόμενη Προεδρία, ότι χρειάζεται επίσημη συζήτηση για έναν αριθμό ε, ζητημάτων σε ό,τι αφορά τις αναπηρίες. Οι διατάξεις ε, περί αναπηριών για την πρόσβαση και την ειδική μεταχείριση των όσων έχουν πληγεί από αναπηρίες. Υπάρχουν εξαιρέσεις για τόπους όπου υπάρχουν συγκεκριμένα πρότυπα για την ε, παρασκευή και την πώληση αγαθών, για την οικοδόμηση νέων κτηρίων, για τις υποδομές, της εγκαταστάσεις και τις μεταφορές. Όλα αυτά πρέπει να συζητηθούν. Και εν τέλει να σας ευχαριστήσω όλους για αυτή την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια οδηγία η Προεδρία γνωρίζει ότι το Ευρωκοινοβούλιο και άλλοι εταίροι επιζητούν χειροπιαστή πρόοδο μετά τις μακροσκελέστατες διαπραγματεύσεις του Συμβουλίου. Όπως όμως προανέφερα και πέραν από τις διάφορες προτάσεις και συστάσει, η Λετωνική Προεδρία θα σε επαφή με πολλά κρατημέλη για να έχει μια σαφέστερη εικόνα για το ποια είναι η τοποθέτησή του για συγκεκριμένα ζητήματα. Ελπίζουμε ότι αυτό θα απασχολήσει και τη Λουξεμβουργιανή Προεδρία για τα διάφορα εκκρεμή ζητήματα. Σα ευχαριστούμε λοιπόν για την προσοχή σα και για την στενή παρακολούθηση αυτού του ζητήματο. Σα ευχαριστώ, Ουλδί και 30 δευτερόλεπτα. Ε, θα προσπαθήσω. για το ποια κράτη-μέλη διστάζουν. Νομίζω τα περισσότερα κράτη-μέλη που στηρίζουν την ε, οδηγία, και είναι πολλά, θα πρέπει να προσπαθήσουν να μεταπίσουν και όσους δεν τη στηρίζουν. Ξέρω ότι κάποιοι ε, είναι επιφυλακτικοί, παρόλο που έχουν ε, εφαρμόσει σχεδόν τα πάντα όσα περιλαμβάνει η οδηγία. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ποιο είναι και το ευρωπαϊκό όφελος, όχι μόνο το ίδιο, και γι' αυτό να εργαστούμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο και ω προς το κόστος Είπατε ότι για όλα τα ζητήματα της προσβασιμότητας, της αναπηρίας, αυτό δεν είναι κάτι που απλώς χρειάζεται να ζητηθεί. Είναι θέμα ίσων δικαιωμάτων και πρόσβασης. Και το ίδιο για τους ανθρώπους με τις αναπηρίες. όπου είναι αυτονόητο δικαίωμα της ανθρώπινης φύσης τους. Διότι Φυσικά και αν αυτοί οι άνθρωποι χάνουν δικαιώματα από τη σκοπιά τη οικονομία και τη αγορά, και παρόλο που δεν μου αρέσει αυτό το επιχείρημα, ναι, χάνουμε και οικονομικά ωφέλη. Πρέπει να δούμε και το κόστο. Έγινε λοιπόν μια μικρή μελέτη για το αντίκτυπο τη μη υλοποίηση αυτών των κανόνων στι μικρομεσαίε επιχειρήσει, αλλά δεν αρκεί αυτό. Τι κοστίζει εάν η οδηγία δεν υλοποιηθεί. Αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε τα κάτι μέλη που επιφυλάσσονται να το λάβουν υπόψη και ε, για αυτό που είπε ο κ. Κυρκόπ για το αν υπήρξε πρόοδος ε, από τη σκοπιά της εκπαίδευσης. Βεβαίως η ευαισθητοποίηση και η αλλαγή της νοοτροπίας είναι κάτι πολύ σημαντικό, αλλά πώς για το γυνατήσιο προσανατολισμό να θυμίσω σε όλους ότι Είχε οδικό χάρτη το Κοινοβούλιο για την ομοφοβία που σκοπό έχει ακριβώς να αλλάξει την οτροπία των ανθρώπων. Και κάτι τελευταίο. Νομίζω ότι η άσκηση πίεσης, και αυτός είναι ο όρος που χρησιμοποιούμε, ε, για να προχωρήσουν τα κράτη-μέλη ε, είναι κάτι που πρέπει να το κάνουμε όλοι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγώ και εσείς και πρέπει να υπάρξει πρόοδος. Αυτό το βλέπουμε ε, και σε νότατα κλιμάκια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζω και ο κύριο Γιούνκερ και ο κύριο Τίμερμαν να μιλάνε στα κρατημέλη που δεν έχουν πιστεί, προσπαθώντα να του πείσουν. Είναι στιγμή να προχωρήσουμε και η οδηγία επιτέλου να γίνει νόμο στα κρατημέλη. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε. Πολύ επί τη ουσία συζήτηση για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ την Προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ και του συναδέλφου. Έρχομαι σε κάτι που κάνει τη δουλειά μου επικίνδυνη και ενθουσιώδη. Θα εξετάσουμε το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Πρέπει να αποφασίσω να δώσω το λόγο στη Σεσίλια και στη Κατερίνα και να κάνω τους υπουργούς να περιμένουν ή να διαγράψω το θέμα από την ημερήσια διάταξη. Σεσίλια, θέλω να είσαι σύντομη. Ναι, για την οδηγία για τους φοιτητές και τους ερευνητές. Τρεις τριμερείς διαλόγους έχουμε κάνει, αλλά χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε τα βασικά πολιτικά ζητήματα. Γίνεται λόγος για τον όγκο των εισδοχών, των εισαγωγών, διαφωνία για τα τεστ για την αγορά εργασίας, για την ενδοευρωπαϊκή κινητικότητα η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο θέλουν αυτά να υπογραμμιστούν. Δεν το στηρίζει αυτό το Συμβούλιο. Συμφωνήσαμε όμως να γεφυρώσουμε τις διαφορές και τα μέλη της οικογένειας. Είναι σημαντική αυτή η οδηγία και έχουμε ένα πνεύμα εργασίας επικοδομητικό. Ευχαριστώ τη Λετωνική Προεδρία για την προσπάθειά της. Προσπάθησε αλλά δεν κατάφερε πολλά. Την ευχαριστώ για την προσπάθεια. Πρέπει να διατηρήσουμε αυτό το πνεύμα εργασίας και να καλωσορίσουμε τη Λουξεμβούργια Προεδρία και να ελπίζουμε ότι αυτή ε, θα τα πάει καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Σεσίλια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήθελε να σχολιάσει για τους φοιτητές και την έρευνα το θέμα, αλλά δεν θέλω να καθυστερούμε. Είναι σημαντικό να μην παρεκκλίνουμε από το χρόνο μας. Θέλω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή... Ξέρω μάλλον ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να πάρει το λόγο και θέλω και εγώ να της δώσω το λόγο, αλλά εν πάση Αλλά δεν υπάρχει χρόνος. Παρακαλώ, ένα λεπτό έχετε, αν μπορείτε σε ένα λεπτό, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα, προσπαθώ, θα προσπαθήσω να είμαι συνοπτικότατη. Την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο είχαμε τον τρίτο τριμερή διάλογο για τις εγγυήσεις ε, δικονομικέ εγγύσει για τα παιδιά που είναι υποπτή κατηγορούμενα στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών. Καταφέραμε συμφωνίες από όλα άρθρα χάρη στην ε, αποτελεσματική συνεργασία τη Λετωνική Προεδρία και τον κομπρεύμα που έδειξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Του ευχαριστώ λοιπόν όλου και του και όλου με του οποίου ήδη βρισκόμασταν σε επαφή κατά την προετοιμασία του τριμερού διαλόγου. Ω προ τα άρθρα για τα οποία πετέχει συμφωνία, πολύ σύντομα να θυμίσω το άρθρο 3, βάσει το το Συμβούλιο δέχτηκε τη θέση του Κοινοβουλίου, όπου σε περίπτωση που υπάρχει αμφιβολία για το ανήλικον ε, ενός για την ηλικία ενός παιδιού θα πρέπει να υπάρχει η απόδειξη δαιμονίας. Έπειτα, για τις διαδικασίες που αφορούν ε, ανηλίκους, θεωρήσαμε ότι η ε, ελευθερία θρησκευτικών πεπιθήσεων και ούτω καθεξής πρέπει να γίνονται σεβαστές όπως αρχικά προβλεπόταν στην οδηγία. Ελπίζω ότι με ικανοποίηση μπορώ να πω ότι αποσπάσαμε οι ανήλικοι κατά τι ποινικέ διαδικασίε και παρόντες να είναι και να μπορούν να συμμετέχουν πλήρω στην όλη διαδικασία και να εκφράζουν και την άποψή του. Και σε αυτή την περίπτωση ε, υπήρξε διεύρυνση τη ε, εγγύηση ε, τη παροχή συνηγόρου, όπω σε υπεράσπιση δηλαδή, ε, σε σχέση με αυτό που προβλεπόταν στην αρχική πρόταση τη Επιτροπή. Βέβαια πρέπει να υπάρξει συνοδεία ενό ενηλίκου και κάποιε άλλε προποθέσει. Παραμένουν ακόμη κάποια σημεία, κάποιε εγγυήσει όπου οι θέσει είναι κάπω διαφορετικέ μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Αλλά πιστεύω ότι στον επόμενο τριμερή διάλογο που θα οργανωθεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα επιληξούμε για Προεδρία, ότι τότε θα έχουμε τη δυνατότητα να καταλήξουμε σε μια καλή συμβαστική λύση. Και βεβαίω θα φροντίσω να ενημερώνω του συναδέλφου τη Επιτροπή. Ευχαριστώ. Thank you, Katerina, Ευχαριστώ, Κατερίνα και συνάδελφοι, διότι με βοηθάτε να διατρέξω επικοδομητικά την ημερήσια διάταξη. Πριν έρθουμε στο σημείο 16, τα συμπεράσματα της Λετωνικής Προεδρίας στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, να σας πω ότι έχουμε τον Υπουργό Εσωτερικών της ε, Λετωνικής Προεδρίας και τον Υπουργό Δικαιοσύνη. Σας καλωσορίζω και τους δύο. Είναι πολύ ενδιαφέρον ε, το ότι είστε εδώ. Θα μπορέσουμε να ακούσουμε τα, συμπεράσματα για, τα συμπεράσματα για αυτό το εξάμεινο. Δεν έχουμε πολύ χρόνο και γι' αυτό δεν θα σας κουράσω με τις εισαγωγικές μου παρατηρήσεις. Σας ζητώ να πάρετε το λόγο μέσω εάν ε, είστε έτοιμοι. Καταρχάς ε, ε, στρέφουμε στον κύριο Κοσλόφσκι, Ρίχαρτ Κοσλόφσκι, Υπουργό Ισοτορικών της Λετωνίας. Έχετε 10 λεπτά να μας παρουσιάσετε την αποτίμηση της δουλειάς σας. Καταρχάς προσωπικά να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία σας κύριε Υπουργέ ε, εκτιμούμε ιδιαίτερως το πνεύμα συνεργασίας που επιδείξατε τους τελευταίους έξι μήνες. Σίγουρα οι συνάδελφοι θα έχουν πολλές ερωτήσεις να σας απευθύνουν. Έχετε το λόγο για δέκα λεπτά όμως, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμο μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι μεγάλη τιμή για εμένα το να βρίσκομαι εδώ σήμερα και να μοιράζομαι μαζί σας την πρόοδο της Λετωνικής Προεδρίας τους τελευταίους έξι μήνες, ειδικότερα ε, στο ε, πεδίο των εσωτερικών υποθέσεων. Η συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι απαραίτητο τμήμα της ε, των προτεραιοτήτων της Λετωνικής Προεδρίας και είναι προς το συμφέρον βεβαίως των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Προεδρία μας θα συνόψιζε τη δράση της στον τομέα αυτό ε, κάνοντας ένα βασικό διαχωρισμό μεταξύ α της εσωτερικής ασφάλειας και β της μετανάστευσης τα καθήκοντα που έπρεπε να φέρουμε σε πέρας μέσα σε αυτό το πλαίσιο των δύο αυτών πυλώνων ε, καθορίστηκαν και επηρεάστηκαν από τις εξωτερικές εξελίξεις. Μετά από τις επιθέσεις 7 Ιανουαρίου ε, και μετά από τις τραγικές εξελίξεις στη Μεσόγειο όλη η Ευρώπη ανησύχησε ιδιαίτερως για τα θέματα ασφαλείας και θελήσαμε να βοηθήσουμε έτσι ώστε να υπάρξει ένα σύστημα για την περιεκτική και ολοκληρωμένη διαχείριση των υφιστάμενων και μελλοντικών προκλήσεων στον τομέα της μετανάστευσης. Συμφωνούμε ότι επάνω στο ότι η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι ομοιόμορφη και ο στόχος μας παραμένει απαράλλακτος, δηλαδή η διατήρηση των αξιών και των ελευθεριών μας το να εγγυηθούμε την ασφάλεια στην Ευρώπη είναι κάτι που πρέπει να συμβαδίζει με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Συνεργαζόμαστε, έχουμε ανοιχτό διάλογο για να έχουμε μια Ευρώπη που θα είναι ένας χώρος ελευθερίας, δικαιοσύνης, δημοκρατίας και αν ε, δράσουμε από κοινού θα έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία έτσι ώστε να προσφέρουμε ασφάλεια στους Ευρωπαίους πολίτες. Κυρίες και κύριοι, ήδη τον Ιανουάριο είπα ότι η μεγαλύτερη πρόκληση που υψώνεται μπροστά μας είναι μία σταθερή και προβλέψιμη πολιτική ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων. Ταυτοχρόνως πρέπει να είμαστε σε θέση να δράσουμε ε, και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις τις συγκυριακές. Και γι' αυτό ξεκινώ με τις προκλήσεις τις μεταναστευτικές. Στα τέλη της περασμένης χρονιάς και στις αρχές αυτής της χρονιάς, Το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν αυτά τα πλοία φαντάσματα, τα οποία ε, μας εξέπληξαν. Το γεγονός δηλαδή ότι οι διακινητές. Είναι όλο και πιο δραστήριοι και η πλεονεξία τους δεν γνωρίζει σύνορα και όλο και προσπαθούν να εξαπλωθούν είναι ε, κάτι το οποίο μας εξέπληξε και γι' αυτό ως Προεδρία δράσαμε αμέσως. Ε, στις 20 Απριλίου μαζί με την ύπατη εκπρόσωπο για θέματα εξωτερικής πολιτικής επικεφαλής της ε, σχετικής υπηρεσίας οργανώσαμε ένα ε, ε, Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνη και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συνδρομή όμως ε, της είπα της εκπροσώπου για να σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Με την υπηρεσία εξωτερικής δράσης συντάξαμε έναν οδικό χάρτη και μέτρα που πρέπει να ληφθούν μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Αυτά έγιναν στις 20 Απριλίου και ε, με ιδιαίτερο μέλημα στις επιχειρήσεις για τη διάσωση της ανθρώπινης ε, ζωής. Ήταν εξαιρετικά σημαντικό να ενισχυθεί η δυνατότητα της Frontex δίδοντας πόρους για ε, την, τις δράσεις στη Μεσόγειο, τριπλασιάζοντας τους πόρους για τις δράσεις στη Μεσόγειο. Επίσης, ήταν απαραίτητο και είναι απαραίτητο να καταπολεμήσουμε τις λανθάνουσες αιτίες, τις βασικές αιτίες πρωταρχικές, οι οποίες αναγκάζουν τους ανθρώπους να ξεκινήσουν μια τέτοια μετάβαση, ένα τέτοιο ταξίδι. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να συνεργαζόμαστε με τις τρίτες χώρες, να ενισχύσουμε τη δυνατότητα αυτών των χωρών και την ανάπτυξη αυτών των χωρών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα μέσα Μαΐου παρουσίασε το νέο πρόγραμμα για τη μετανάστευση, βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο, μακροπρόθεσμο. Ε, καθήκοντα και στόχοι δηλαδή σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο για να έχουμε μια νέα ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική. Η Πρόεδρος ξεκίνησε τις συζητήσεις αμέσως, ο Πρόεδρος, και σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι το Συμβούλιο στηρίζει το πρόγραμμα και τα μέτρα που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία εκτείνεται σε τέσσερις πυλώνες. Πρώτον, εξάλληψη της παράνομης παράτυπης μεταναστευτικής ροής. Δεύτερον, ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων. Τρίτον, ε, διόρθωση του συστήματος για, για το άσυλο και τέταρτον, No Legal Migration Policy. Είναι απαραίτητο να διασφαλίσουμε ότι η ευρωπαϊκή πολιτική είναι ισορροπημένη και μεγιστοποιεί τα ωφέλη της νόμιμης μετανάστευσης και δίδει άσυλο σε αυτούς που το αξίζουν. Ενώ ταυτόχρονα καταπολεμάται η παράτυπη ή παράνομη, η legal μετανάστευση. Είναι αποκλίνουσες οι απόψεις για τα μέτρα αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αναδιάχυση των ανθρώπων μέσα στην Ευρώπη, για την ε, κατεύθυνσή τους ε, αλλού μέσα στην Ευρώπη. Συζητήθηκε το θέμα αυτό περίπου για 6 ώρες μεταξύ άλλων, χθες και το Συμβούλιο στα τέλη του Ιουνίου θα είναι καθοριστική σημασίας. Έχουμε κοινή αντίληψη του γεγονότος ότι είναι απαραίτητο να στηρίξουμε τις χώρες που υποφέρουν από πολύ υψηλές μεταναστευτικές πιέσεις. Έχουμε συμφωνήσει σε, πάνω σε διάφορες λεπτομέρειες του μηχανισμού για να έχουμε ένα, μια δίκαιη αντιμετώπιση, fairness. Οι συζητήσεις στο Συμβούλιο θα συνεχιστούν εντατικά για να εξευρεθεί συμβιβαστική λύση. Είναι τώρα σαφές ότι δεν υπάρχει ένα οικουμενικό ενιαίο εργαλείο για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις μεταναστευτικές ροές. Πρέπει να έχουμε αντιθέτως μια συνολική, περιεκτική προσέγγιση, ολοκληρωμένη. Και καλωσορίζουμε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ε, την ε, για την έκθεση αυτή και, και καλωσορίζουμε και την έκθεση του Κοινοβουλίου σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι, οι νόμιμες δίωδοι μετανάστευσης, τα νόμιμα εργαλεία μετανάστευσης είναι καλό τρόπος να διαχειριστούμε τις μεταναστευτικές ροές. Πρέπει να υπάρξει καινή θέση σε σχέση με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για τους ερευνητές και τους φοιτητές. Σίγουρα έχουμε προχωρήσει σε αυτό το πεδίο, αλλά παραμένουν ζητήματα που ε, θα συζητήσουμε εντακτικά για να βρεθεί ε, συμβιβαστική λύση. Ένας επικοδομητικός διάλογος θα μας επιτρέψει να καταλήξουμε σε συμφωνία μέχρι τα τέλη της χρονιάς. Συνεχίζουμε τις εργασίες μας εντατικά ως προς τους στόχους για τις θεωρήσεις, για τις βίζες. Έχουμε κάνει πολλά ώστε τους επόμενους έξι μήνες να μπορέσει να επιτευχθεί συμφωνία εντός Συμβουλίου και έτσι να ξεκινήσει ο διάλογος στη συνέχεια με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις προτάσεις αυτές. Έχουμε φτάσει σε συμφωνία επίσης ως προς τον κανονισμό του Δουβλίνου και τις ε, τροποποιήσεις αυτού. Συζητήσαμε την προστασία των πιο ευπαθών ομάδων και κυρίως των ανηλίκων για να κατανοήσουμε καλύτερα γιατί ο κόσμος επιλέγει να παραβιάσει αυτό που προβλέπεται στη βίζα του ή στην άδεια παραμονής τους, έχουμε ε, την επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Amber Light. Και ήταν απαραίτητο να... Από την 55 ε, θα ήθελα να πω ότι πολλά κράτη-μέλη πήραν μέρος σε αυτή τη ε, δραστηριότητα και συνέλεξαν στοιχεία από 25 αεροδρόμια. Κανείς δεν ε, συνελήφθη παρόλο που φάνηκε ότι τα έγγραφα είχαν λήξει. Από 36 αεροδρόμια λάβαμε 230 τόσες αναφορές, διάβαμε διάφορα στοιχεία για 1003 περίπου ανθρώπους. Όλα αυτά είχαν ερευνητικό σκοπό για να καταλάβουμε περισσότερο τις αιτίες και στην αρχή της χρονιάς ξεκινήσαμε ένα πιλωτικό project για τα έξυπνα σύνορα. Το Συμβούλιο συνέχισε ε, τη δουλειά του για αυτό το έξυπνο πακέτο Smart Border Package και θα είναι η βάση για τη δουλειά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει τη νέα της πρόταση για τα έξυπνα σύνορα. Είναι απαραίτητο να συνεχιστεί όλη αυτή η δουλειά για να αξιοποιήσει κανείς τα ωφέλη της νέας τεχνολογίας. Ταυτοχρόνως πρέπει να έχουμε υπόψη και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Κυρίες και κύριοι, όπως ανέφερα ήδη, η μετανάστευση δεν είναι η μόνη πρόκληση που αντιμετωπίσαμε κατά τη διάρκεια της προεδρίας μας. Ε, μετά τις εξελίξεις και τα γεγονότα στο Βέλγιο, στη Γαλλία και στη Δανία είδαμε ότι η τρομοκρατία ε, αποτελεί μεγάλη ε, πηγή κινδύνου για την ασφάλεια της Ευρώπης. Στις 29 πρώτου στη Ρήγα οι Υπουργοί Εσωτερικών Υποθέσεων συζήτησαν τις προκλήσεις στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Και είμαι ικανοποιημένος διότι το Συμβούλιο Υπουργών κατέληξε στην κοινή δήλωση της Ρήγας, κάτι το οποίο συνέβαλε στην περαιτέρω συζήτηση για την καταπολέμηση του φαινομένου αυτού και ε, ε, έγινε η συζήτηση στην άτυπη σύνοδο κορυφής μετά τις 20 Φεβρουαρίου περίπου. Και θέλουμε να έχουμε ισορροπία μεταξύ των εγγυήσεων για την ασφάλεια από τη μία και της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων από την άλλη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μας έχει ζητήσει να φέρουμε σε σε πέρα σε αυτό το καθήκον, να έχουμε ασφάλεια εγγυήσει για την ασφάλεια και εγγυήσει για το, την προστασία των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και είναι αυτό μια πολύ καλή βάση για να συνεχίσουμε τον αγώνα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Τέσσερις προτεραιότητες είναι αυτές που επιλέξαμε για να ε, προχωρήσουμε και να πετύχουμε καλά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της εξάμηνης προεδρίας μας. αξιοποιήσαμε τις δυνατότητες του πλαισίου Σέγγεν για να ενισχύσουμε και να εξυγχρονίσουμε τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων και να ασχοληθούμε με ε, τον ακραίο εξτρεμισμό και την τρομοκρατία εντός εξωτερικών συνόρων, τη ριζοσπαστικοποίηση, καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου όπλων και λύσεις κατά προτεραιότητα ως προς τον αφοπλισμό από τα πυροβόλα όπλα και την απενεργοποίησή τους. Αυξημένη ανταλλαγή πληροφοριών, ενίσχυση συνεργασίας σε επίπεδο Europol και Eurojust. Όλες αυτές ήταν οι προτεραιότητές μας. Και το κύριο αίτημα ήταν να αναζητήσουμε δυνατότητες πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα διαθέσιμα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας Επετεύχθη πρόοδος, επετεύχθη συμφωνία και σαν αποτέλεσμα την 1η Ιουλίου θα έχουμε μια νέα ομάδα που θα δημιουργηθεί από πλευράς Ευρωπόλ που θα αναφέρεται σε σχέση με τα περιεχόμενα του διαδικτύου για να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τους υφιστάμενους πόρους πιο αποτελεσματικά μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπόλ σχεδιάσαμε να δημιουργηθεί ένα κέντρο κατά της τρομοκρατίας ε, εντός της Ευρωπόλ. Ταυτόχρονα θα πρέπει να ομολογήσω ότι το φαινόμενο των ξένων των αλλοδαπών μαχητών παραμένει μία από τις μεγαλύτερες απειλές ε, στην ασφάλειά μας, εσωτερική ασφάλεια και πρέπει να εξεύρουμε τρόπους πώς θα αντιμετωπίσουμε και θα εξουδετερώσουμε αυτή την απειλή. Δεύτερον, πρέπει να αξιολογηθούν οι δυνατότητες να βελτιωθεί η νομοθεσία μας, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου ο στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί διαφορετικά, με διαφορετικά μέσα. Ένα από τα πεδία όπου ήταν αναγκαίες τέτοιες ε, αλλαγές ε, ήταν η αντιμετώπιση των ε, παράνομων πυρομαχικών και υλικών και η πρόταση για ένα νομοθετικό πλαίσιο όπως θα ήταν δυνατόν να υποβληθεί το δυνατόν ταχύτερα. Το Συμβούλιο με θετικό τρόπο ε, αντιμετωπίζει τις δραστηριότητες ε, του Ευρωκοινοβουλίου σε σχέση με την διαβίβαση προσωπικών δεδομένων ταξιδιωτών ώστε να υπάρξει ένας μηχανισμός ε, για την επεξεργασία τέτοιων δεδομένων. Το Συμβούλιο θεωρεί ότι αυτό είναι ένα αποτελεσματικό θεμελιώδους σημασίας μέσο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Χρειαζόμαστε έναν αποτελεσματικό μηχανισμό που θα σέβεται τις ε, διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων αλλά θα είναι και αποτελεσματικός όσον αφορά την ασφάλεια. Θετικά διάκυμε έναντι του διαλόγου, ανοιχτού διαλόγου και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να εξεύρουμε συμβιβαστικές λύσεις και ευελπιστώ ότι και οι δύο συνομοθέτες θα μπορέσουν να εξεύρουν μια λύση με μια συμφωνία πριν από τα τέλη του έτους. Όπως προανέφερα ήδη τον Ιανουάριο, θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα ωφέλη τα οποία θα μπορούσαν να δοθούν από μια τέτοια διαδικασία για την καταπολέμηση των απειλών. Οι απειλές από την τρομοκρατία όμως δεν είναι οι μόνες απειλές που αντιμετωπίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εργαστήκαμε πολύ έντονα σε βάθος κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών με τη, για την στρατηγική, την εσωτερική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εχθές κατά την συνάντηση συμφώνησαν οι Υπουργοί σε ένα πλαίσιο για αυτή την εσωτερική στρατηγική για τα επόμενα πέντε χρόνια καθορίζοντας, θεσπίζοντας προτεραιότητες και καθορίζοντας επίσης τους τρόπους ε, εφαρμογής, ε, υλοποίησης και εποπτείας. Η κύρια πρόκληση είναι να μπορέσουμε στην πρακτική εφαρμογή να υλοποιήσουμε όλα αυτά τα οποία συμφωνήθηκαν. Γι' αυτό πρέπει να αναπτυχθούν και να καταρτιστούν τα αναγκαία έγγραφα για την εφαρμογή και υλοποίηση όλων αυτών. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας εργαστήκαμε έντονα για να καταλήξουμε σε συμφωνίες ε, όσον αφορά τις ε, διαδικασίες ε, Seaboard και Europol. Χάρη στη συνεργασία ακριβώς με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με την εισηγήτρια καταφέραμε να επιτύχουμε πρόοδο σε αυτό το χαρτοφυλάκιο. Όμως πιστεύουμε ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στην εξέβρεση μιας επικοδομητικής συμφωνίας. Όσον αφορά τον κανονισμό Europol υπάρχουν κάποια θέματα που εκκρεμούν, κάποια ανοιχτά ερωτήματα. Όμως ευελπιστούμε ότι στον διάλογο με ε, τον συγητή υπάρχει μια θετική βάση για την επίτευξη συμφωνίας κατά τη διάρκεια του επόμενου εξαμήνου. Θα ήθελα αν επιτρέπετε τώρα να στραφώ στην εξωτερική διάσταση αυτών των θεμάτων. Η εξωτερική αυτή παράμετρος επηρεάζει τα θέματα της εσωτερικής ασφάλειας, διότι οι μεταναστευτικές ροές και η εσωτερική ασφάλεια συνδέονται και εξαρτώνται από εξωτερικά γεγονότα. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε εξάλλου, η προτεραιότητά μας ήταν συνεργασία με τις χώρες εταίρους της Ανατολικής Γειτονίας και σε υπουργικές συναντήσεις, ε, οι συναντήσεις Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων Δικαιοσύνης ε, ε, έλαβαν χώρα όπου συζητήσαμε την ενδυνάμωση του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δημοκρατίας. Αυτά τα θέματα συζητήθηκαν και μέσα στο πλαίσιο της προσπάθειας καταπολέμησης της διαφθοράς. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας δώσαμε ιδιαίτερη προσοχή στην ενδυνάμωση της συνεργασίας με την Λευκορωσία Μπέλαρους και με χαρά μπορούμε να αναφέρουμε ότι υλοποιούνται οι διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2014 ενώ η επίσημη υπογραφή ακυρώθηκε κατά την τελευταία στιγμή λόγω τεχνικών λόγων, η κοινή διακήρυξη όσον αφορά την ε, εταιρική αυτή σχέση μέσα στο πλαίσιο της γειτονίας με την Πέρα υπογραμμίστηκε. η υψηλή αξιωματούχοι μετά από τις πρώτες επαφές ε, διαπιστώνουν ότι υπάρχει πρόοδος που επετεύχθη σε όλους τους τομείς. Θέλω να ευχαριστήσω για αυτή την επικοδομητική αντιμετώπιση. Μόνο με στενή συνεργασία μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους μας, να διασφαλίσουμε τα, την Ευρώπη και να είναι σεβαστά τα δικαιώματα του ανθρώπου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα ο Υπουργό Δικαιοσύνη θα λάβει τον λόγο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κυρίες και κύριοι, χαρά είναι για μένα να παρίσταμαι εδώ σήμερα ενώπιόν σας για να συμμεριστώ μαζί σας τις πρόοδους που επετέφθησαν από την Λετωνική Προεδρία στον τομέα της δικαιοσύνης. Θα συνεχίσω τώρα τον λόγο μου στην λετωνική γλώσσα. Ένα από τα κύρια θέματα και στόχους της Λετωνικής Προεδρίας ήταν και είναι η διασφάλιση των στόχων της ε, Προεδρίας και η συνέχιση της εργασίας στο Συμβούλιο που ξεκίνησε υπό την Ιταλική Προεδρία κατά το πρόσφατο παρελθόν. Εργαζόμαστε και εργαστήκαμε έντονα ώστε να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Προτού παραδώσουμε τη σκητάλη της Προεδρίας στο Λουξεμβούργο ως επόμενη Προεδρία σε, μετά από δύο εβδομάδες κατά την 1η Ιουλίου Αυτά που μπορούμε να πούμε είναι ότι κατά την έναρξη της Προεδρίας μας σας ενημερώσαμε για τις προτεραιότητες της Λετωνικής Προεδρίας στον τομέα της δικαιοσύνης. Και αυτές οι προτεραιότητες ε, εξάλλου εντάσσονται στο πλαίσιο των στόχων της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών ΛΥΜΠΕ της, ε, ε, της Ευρωβουλής ενίσχυση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, προστασία των χρηματοοικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενδυνάμωση των δικαιωμάτων των υπόπτων και των κατηγορουμένων στην ποινική δικαιοσύνη, καθώς επίσης και η περαιτέρω ανάπτυξη της έννοιας δικαιοσύνη για την ανάπτυξη, justice for growth έχοντας συνειδητοποιήσει ότι η προστασία των δεδομένων βρίσκεται πάνω-πάνω ε, στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Λετωνική Προεδρία θεώρησε αυτόν τον στόχο και τον καθόρισε ως έναν από τους κυριότερους στόχους της Προεδρίας της. Από κοινού με συναδέλφους άλλων κρατών μελών καταβάλαμε μέγιστες προσπάθειες για την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων στην προστασία των δεδομένων και στέφθηκαν με επιτυχία αυτά τα, αυτές οι προσπάθειες. Καταλήξαμε μετά από διαβουλεύσεις ε, που συνεχιζόντουσαν επί περισσότερο από τρία έτη σε συγκεκριμένα από τα χειροπιαστά αποτελέσματα. Και για να καταφέρουμε να επιτελέσουμε το έργο μας με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για την μεταρρύθμιση, την αναθεώρηση της προστασίας των δεδομένων, ξεκινήσαμε με μια γενική προσέγγιση κανονισμού για την προστασία των δεδομένων. Και κατά τη διάρκεια της εξάμηνης προεδρίας μας επιτύχαμε θετικά, επικοδομητικά αποτελέσματα με τιμά το ότι μπορώ να αναφέρω ότι κατά την 15η Ιουνίου στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης πετύχαμε καταφέραμε να καταλήξουμε σε μια γενική συμφωνία επί του κειμένου του κανονισμού αυτού. Αυτό θα μας επιτρέψει όχι μόνο να ξεκινήσουμε τον τριμερή διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά επίσης θα μας δώσει την ευκαιρία και την δυνατότητα να ολοκληρώσουμε, να ολοκληρώσουμε το έργο μας όσον αφορά την οδηγία για την προστασία των δεδομένων το δυνατόν ταχύτερα. Είμαι ευγνώμων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ευκαιρία που μας παρήχε να ξεκινήσει η διαδικασία των τριμερών διαλόγων ήδη κατά την 24η Ιουνίου. Μπορούμε να πούμε ότι με την έγκριση αυτή της προστασίας δεδομένων από το Συμβούλιο έχουμε ένα σημαντικό γεγονός ε, ενώπιόν μας, μεγάλης εμβέλειας και μπορούμε να ολοκληρώσουμε την Προεδρία μας ε, με ικανοποίηση ε, λόγω αυτού. Όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προτεραιότητα της Λετωνικής Προεδρίας είναι ο κανονισμός για την θέσπιση της ε, επίτευξης της ε, Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ως θεσμού. Συνεχίζουμε το έργο που προηγήθηκε από προηγούμενες προεδρίες. Έχοντας ολοκληρώσει το έργο επιβασικών αρχών για αυτό το θέμα, για τα πρώτα άρθρα του ε, κανονισμού για την εισαγγελία, στην αρχή κατά την έναρξη της Προεδρίας μας είχαμε και έντονες συζητήσεις όσον αφορά τα θέματα που εκκρεμούσαν και δεν είχαν ακόμη ρυθμιστεί. Κατά τη Σύνοδο του Μαρτίου των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων συζητήσαμε τον καθορισμό, τον, ε, τη δημιουργία της ε, Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τις δομές που θα έχει και την δυνατότητα ε, ακριβώς διορισμού ε, στελεχών σε αυτή την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Παρότι είναι ιδιαίτερα περίπλοκα και σύνθετα όλα τα ζητήματα, σημειώσαμε σημαντική πρόοδο και παρόλα αυτά μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει πολύ έργο που πρέπει ακόμη να επιτελεστεί και που απομένει να γίνει. Η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα είναι ένα από τα δυσχερέστερα ε, εγχειρήματα ως πρόκληση της ε, Λουξεμβουργιανής Προεδρίας. Τρίτον, για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τους προηγούμενους έξι μήνες ε, εργαστήκαμε για την οδηγία επί για την καταπολέμηση της διαφθοράς ε, και των απατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την πέμπτη οδηγία. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι επετεύχθη συμβιβασμό επί κάποιου αριθμού θεμάτων, ιδιαίτερα για τη συμπερίληψη και της ε, απάτης όσον αφορά τον ΦΠΑ, που είναι εξίσου σημαντική υπόθεση και για το Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Οι πραγματογνώμονες μας, οι εμπειρογνώμονες εργάστηκαν και για την ομοθεσία Eurojust που ε, στοχεύει στο να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της Eurojust δημιουργώντας ένα νέο πρότυπο <clears throat> διαχείρισης και διακυβέρνησης και βελτιώνοντας την λειτουργική αποτελεσματικότητα μέσω ενός ενιαίου ορισμού <clears throat> των αρμοδιοτήτων και του καταστατικού και καθεστώτος των εκπροσώπων. Επίσης ε, για την επίτευξη μιας γενικής συμφωνίας κατά το Μάθιο από πλευράς των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων οι στόχοι επετεύχθησαν. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα το οποίο μας απασχόλησε ήταν η ενίσχυση, ήταν ακριβώς ε, η ενδυνάμωση του θέματος των δικαιωμάτων όσον αφορά τους υπόπτους και τους κατηγορούμενους στην ποινική, ε, στην ποινική διαδικασία, ε, ποινική δικαιοσύνη. Ε, όσον αφορά την επίτευξη ενός δεσ... μιας δέσμης μέτρων για την νομική αρρωγή και υποστήριξη. Στόχος ήταν ο καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών για την ενδυνάμωση των δικαιωμάτων των κατηγορουμένων και υπόπτων στην ποινική δικονομία ε, και όσον αφορά τις επαφές ε, πραγματογνωμόνων ε, με κοινέ προσπάθειες καταλήξαμε σε μια συμφωνία επ' του χαρτοφυλακίου και κατά τον Μάρτιο ήδη τη, μεταξύ Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων για τα άλλα δύο χαρτοφυλάκια, δηλαδή για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών και ανηλίκων και την ε, προστασία των ε, ε, κατηγορουμένων. Εργάστηκαν έντονα οι εμπλεκόμενοι για να επιτευχθεί η μέγιστη πρόοδος όσον αφορά την έγκριση αυτών των δύο χαρτοφυλακίων. Ταυτόχρονα θα ήθελα να τονίσω ότι δεν πρέπει να καθυστερήσουμε πλέον την έγκριση αυτών των χαρτοφυλακίων ιδιαίτερα του χαρτοφυλακίου των δικαιωμάτων των παιδιών διότι τα παιδιά είναι μία από τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και πρέπει να προστατεύονται φυσικά. Ολοκληρώνοντας θα ήθελα θερμά να ευχαριστήσω την ομάδα που με βοήθησε, που με τόση ζωτικότητα και τις ικανότητες και δεξιότητες ε, με ε, βοήθησε και με υποστήριξε. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης ε, τους Ευρωβουλευτές μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, ΛΥΜΠΕ της Ευρωβουλής, ε, για την εμπιστοσύνη τους. Ήταν πραγματικά ιδιαίτερη χαρά να έχω συνεργαστεί μαζί σας κατά τους έξι μήνες. Um, Ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσουμε με τους συντονιστές. Ε, θέλετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να εκφράσω τη βαθιά μου εκτίμηση σε αυτά που είπε ο κύριος Κοσλόφσκης ως προς τη μετανάστευση. Να πω ότι πρέπει όλες τις πτυχές του θέματος να τις δουλέψουμε. Όμως στη δημόσια συζήτηση μιλούμε μόνο για την καταπολέμηση των διακινητών για τις ποινικέ διώξεις, για, το σύνολο των, για τον έλεγχο των συνόρων μας, για τη δημιουργία στρατοπέδων χωρίς καν να ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Άρα η εντύπωση που δίνουμε ως Ευρώπη είναι ότι δεν θέλουμε να έχουμε μετανάστες. Και αυτό υπογραμμίζεται από το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν ήταν σε θέση να ε, καταλήξει σε μία απόφαση για την κλίδα κατανομής και προώθησης μεταναστών μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μου απαντήσετε σε αυτό το ερώτημα, όμως σας ρωτώ ποια είναι τα κράτη-μέλη που στήριξαν ξεκάθαρα την ιδέα της επανεγκατάστασης ή ανατοποθέτησης, relocation, ή να μας πείτε τουλάχιστον πόσα κράτη-μέλη είναι υπέρ του relocation και του προγράμματος επανα ή αναεγκατάστασης, resettlement, ή όλοι έχουν πρόβλημα με αυτό. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι όλα τα κράτη-μέλη χρειάζονται τη μετανάστευση στη Γερμανία χρειαζόμαστε 300.000 μετανάστες σε διάφορους τομείς της εργασίας μας τα επόμενα χρόνια. Όμως δεν υπάρχει ευρωπαϊκός κανόνας για τη μετανάστευση πέρα από την μπλε κάρτα. Νομίζω ότι σε κάθε χώρα χρειάζονται μετανάστες σε διάφορους τομείς προσόντων και είναι έτοιμα τα κράτη-μέλη για να συνεργαστούν ε, με τους κλάδους της οικονομίας. Από εκεί και πέρα, για το τομέα της προστασίας των δεδομένων, στρέφομαι στον Υπουργό Δικαιοσύνης για να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Ράσναστ. Θα έχουμε οδηγία, ελπίζουμε, τον Οκτώβριο για το κοινοβουλίο το πακέτο, οι δέσμοι μέτρων για την προστασία των δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντικό. Θέλω να μας πείτε περισσότερα για αυτό. Τώρα για τις οικονομικές εγγυήσεις για τους υπόδικους ανηλίκους, πράγματι πολλή δουλειά έχει γίνει και ελπίζουμε ε, το εφαλτήριο που δόθηκε με τη δική σας Προεδρία να οδηγήσει ε, στο κλείσιμο της υπόθεσης και με το τέλος της επόμενης Προεδρίας. Ευχαριστώ. δεν θα κάνω εγώ ερώτηση που να είναι ανεξάρτητη, αλλά θα συμπληρώσω μια ερώτηση των όσων είπε η Μπίργκιτ για το Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων και την έλλειψη συμφωνίας. Να ρωτήσω, μια και επικεντρώθηκε η ερώτησή της στις χώρες. Ξέρουμε ότι δεν υπήρξε συμφωνία και ο Επίτροπος Αβραμόπουλος ήταν ουδέτερος στα σχολεία του. Τι πρόπτικη υπάρχει κατά την άποψή σας μια και τελειώνει η Προεδρία σα να επιτευχθεί συμφωνία τον Ιούνιο, τον Ιούλιο. Έχετε ελπίδε ότι μπορεί να συμβεί αυτό. Και μιας και έρχεται στο τέλος του εξαμήνου. Οι χώρες που γνωρίζουν ιδιαίτερη πίεση, τι θα κάνουν εφόσον δεν υπάρχει συμφωνία. Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει αλληλεγγύη σε αυτού του είδου Θα ήθελα λοιπόν να συμπληρώσω την ερώτηση της συναδέλφου και να μου πείτε αν ε, έχετε κάποια άποψη για τους συντηρικούς μεταρρυθμιστές, ο κύριος Κύρκο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να συγχαρώ την Προεδρία για τη δουλειά του. Νομίζω ότι πραγματικά ήταν ε, πολύ δραστηρή από τις πληροφορίες μου. Γνωρίζω ότι σε πολλού τομεί και ιδιαίτερω σε αυτόν πέτυχαν πάρα πολλά αποτελέσματα για το διάρκεια της προεδρίας τους. Έχω όμως δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις παρακαλώ. Κατά πρώτον, επειδή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που τα κάτι μέλη φαίνεται να ανταγωνίζονται για τις θεωρήσεις που απειλούν να εκδώσουν κράτη-μέλη ε, εναντίον όσων δεν συνεργάζονται στα θέματα του αναπατρισμού, τη επιστροφή και το καθεξή. Πιστεύει η Προεδρία ότι η θεώρηση και η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους υποχρεωτικούς κανόνες μπορούν να υλοποιηθούν. Και αν ναι, σε τι βαθμό. Και σε ποιο χρονικό πλαίσιο. Το θέμα αυτό με ενοχλεί ιδιαίτερως αυτή τη στιγμή. Ε, και επίσης η Προεδρία θεωρεί ως προς τα σύνορα ότι τα ευφύ σύνορα και οι σχετικοί θέσμοι μέτρων είναι ένα σημαντικό στοιχείο για την νέα ε, πολιτική θεωρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές προτάσεις. Ιδίως μια πρόταση που έχει γίνει από κάποιους, το πεδίο των αρχικών προτάσεων να διευρυνθεί. Προφανώς, ε, εγώ πιστεύω, όπως έχει υποθεί και προηγουμένως, δεν ξέρω τι πιστεύετε εσείς, ότι η νόμιμη μετανάστευση η οικονομική μετανάστευση και το άσυλο είναι θέματα που πρέπει να τα βλέπουμε με κάποια συμπάθεια μεν, με θετικό τρόπο, αλλά αυτόνομα. Τι άποψη λοιπόν έχει το Συμβούλιο για την ε, διάθεση κάποιων κρατών μελών να έχουν ένα ευρύτερο πεδίο, ένα ευρύτερο φάσμα διοικητικών μέτρων για να καλύπτουν τις διαφορές μεταξύ αυτών των διαφορετικών στοιχείων. Και σε αυτή τη φάση να ευχαριστήσω και την Προεδρία ιδιαιτέρω για τη στήριξη και τη συνδρομή του προ εμένα για το Μητρό Επιβατών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και την όλη διαδικασία για το οποίο υπήρξε εισηγητή. Δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά ε, για τη διάρκεια τη Προεδρία του του ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία. Και επίση να ρωτήσω ε, την Προεδρία για την εξέλιξη της τρομοκρατικής μονάδας στην Europol. Πώς το βλέπετε αυτό, ιδίως ε, λόγω των ευαισθησιών που υπάρχουν ένθεν και ένθεν για τη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις εθνικές αρμοδιότητες σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστούμε για τους φιλελευθέρους, κυρία Βίκστρομ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί Υπουργοί, Νομίζω οφείλω να σας συγχαρώ για την πρώτη σας ε, προεδρία που σύντομα θα ολοκληρωθεί. Νομίζω ότι η δουλειά που είχατε ήταν πραγματικά άφθονη. Όχι μόνο για να αποκριθείτε στις δημοκρατικές επιθέσεις και τις απειλές στην αρχή της Προεδρίας σας, αλλά και για τα υπόλοιπα. Μπράβο σας λοιπόν, σταθήκατε στο των περιστάσεων και ευχαριστούμε για τις σημερινές σας ομιλίες. Έχω κάποιες ερωτήσεις Έχουμε συνεργαστεί στενά για τους φοιτητές, τους ερευνητές και το σχετικό φάκελο. Είναι καλό που ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσει και μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε τρει γύρου τριμερών διαλόγων. Όμως, λυπούμε που δεν καταφέραμε να ε, έχουμε ουσιαστικότερη πολιτική πρόοδο για το θέμα αυτό. Είναι τόσο πολλά τα εκκρεμή ζητήματα που ε, θα πρέπει να τα επιλύσουμε τις ερχόμενες ημέρες, αλλά δεν μπορώ παρά να ευχαριστήσω για τις προσπάθειές σας. Τις τελευταίες εβδομάδες ιδιαιτέρως ελπίζω ότι θα έχετε την τόλμη να πείτε στα υπόλοιπα ότι τώρα επιτέλους πρέπει να προχωρήσουμε λίγο, εάν θέλουμε ανταγωνιστικότητα και να είμαστε και ελκυστικοί για τους ε, λαμπρότερους εγκεφάλους, τους καλύτερους φοιτητές και ερευνητές που τόσα απεγνωσμένα χρειαζόμαστε σε αυτή την Ήπειρο για να έχουμε ευημερία και στο μέλλον. Ελπίζω ότι εάν έχουμε όλη την ίδια σοβαρή προσέγγιση θα πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτό το φάκελο. Αυτό θα πρέπει να είναι η μαρτυρία σας για την Λουξεμβουργιανή Προεδρία που θα αναλάβει τώρα. Όσο αφορά την τραγική κατάσταση στη Μεσόγειο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα με συγκεκριμένα μέτρα. Εμείς από το σώμα αυτό είμαστε πολύ σαφείς στο ψήφισμα που εγκρίναμε τον Απρίλιο για το πού θέλουμε να οδεύσουμε από πολιτικής σκοπιάς. Δύο θεσμικά όργανα λοιπόν είναι βαθιά πεπισμένα ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι ανάληψη ευθύνης και κατανομή των ευθυνών Καλό θα ήταν να περάσουμε από την κατανομή όπως ονομάζεται του άχθους, burden στην κατανομή και την ε, κοινή ανάληψη ευθύνη. Διότι τα ανθρώπινα όντα δεν μπορεί να θεωρούνται άχθο και βάρο. Ε, έχουμε πετύχει λοιπόν πολλά. Ε, το πνεύμα ήταν θετικό, όμω πρέπει να υπάρξει πρόοδο στα κράτη-μέλη πλέον. Η αρχική απόκριση των κρατών μελών δεν ήταν πολύ θετική, για να μην το πω διαφορετικά μάλλον το αντίθετο, αλλά βλέπουμε ακόμη και σήμερα διμερείς συγκρούσεις, τις οποίες ε, τις πυροδοτούν τα κράτη-μέλη που απειλούν να κλείσουν τα σύνορά τους, να ενεργήσουν ακόμη πιο περιοριστικά. Ελπίζω ότι πραγματικά θα εκμεταλλευτείτε τις τελευταίες μέρες της Προεδρίας σας για να διευκολύνετε και να εξομαλύνετε αυτές τις διαφωνίες, για να κινηθούμε στη σωστή κατεύθυνση και να βεβαιωθούμε ότι εν τέλει θα μπορέσουμε να υιοθετήσουμε συγκεκριμένα μέτρα και όχι μόνο να μείνουμε στα λόγια. Ε, ωραία είναι η φλιαρία, αλλά την Κυριακή λέμε ένα πράγμα και τη Δευτέρα το πρωί το αντίθετο. Βλέπουμε τρομακτικές δράσεις από τα κρατη Μας τρομάζουν. Και να επιστρέψω σε αυτό το που είπε ο συνάδελφος, ε, Θέλουμε να ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που εκφράζουν αυτές τις απόψεις και τι ακριβώ λένε για να μπορέσουμε να ασκήσουμε πίεση. Για τον κανονισμό του Δουβλίνου, όπου είμαι εισηγητρία, είναι ξεκάθαρη περίπτωση. Υπάρχει απόφαση του δικαστηρίου για το πώ θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε στου ασυνόδευτου ανηλίκου. Και η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι απλούστατα να ε, μεταφέρουμε την απόφαση του δικαστηρίου σε νομοθέτημα, να τη μεταφράσουμε σε νομοθέτημα. Ένα θέμα είναι με ένα άρθρο. Τα κράτη-μέλη του δίνουν τρομακτικέ διαστάσει, προσπαθούν να βρουν εναλλακτικέ ερμηνείε. Δεν υπάρχει ε, συζήτηση επί τη ουσία γι' αυτό. Σε αυτό το σώμα έχω την πλήρη στήριξη όλων. Δεν υπήρξε καμία τροπολογία για το θέμα. Θα πρέπει απλώ να το καταπιούν στο Συμβούλιο και θα πρέπει να περάσετε το μήνυμα και στους υπολείπους. Για την προστασία των δεδομένων, βεβαίως καλώς ορίζουμε την πρόοδο που έχει επιτελεστεί, ιδίως αυτή την εβδομάδα. Τη Δευτέρα ελπίζουμε ότι θα υπάρξει ένα φιλόδοξο αποτέλεσμα για όλο το πακέτο και δεν θα συμφωνήσουμε με διατάξεις που δεν θα παραμείνουν στα πρότυπα της οδηγίας του 95. Τώρα, πώς προβλέπετε να εξελιχθεί η οδηγία αυτή και η έγκρισή της. Είναι ζωτική σημασία αυτό. Και η τελευταία μου ερώτηση είναι η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδίω στην Ουγγαρία. Την τελευταία εβδομάδα το Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα απολύτω ξεκάθαρο ψήφισμα, όπου εκφράζει τη φλήψη του για την έλλειψη αντίδραση από το Συμβούλιο προ τι πολυάριθμε ανησυχητικέ εξελίξει του τελευταίου διαστήματο στην Ουγγαρία κατά τη διάρκεια τη Προεδρία σα. Θανατική ποινή διακριτική μεταχείριση μεταναστών. Αυτά ανακύπτουν διαρκώς. Θα μπορούσα να επεκταθώ. Ε, και επίσης φήμες από την Προεδρία ότι δεν συζητήθηκε μια φορά. Έτσι είναι. Και πώς θα το δικαιολογούσατε. Γιατί δεν υπήρξε κανένας διάλογος για το θέμα αυτό. Μια συζήτηση. Επίσης ήθελα τη γνώμη σας για έναν βαθμιαίο και μη δεσμευτικό μηχανισμό ώστε να βεβαιωθούμε ότι τα κριτήρια της Κοπενχάγης ε, εκπληρώνονται από τα κάτι μέλη εφόσον είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήταν ενδιαφέρον να το ξέρουμε και αυτό. Σας ευχαριστώ και καλή διασκέδαση στις τελευταίες εβδομάδες της Προεδρίας σας. Ευχαριστούμε, Σεσίλια. Μίλησε σαν να ήσουν Υπουργός Δικαιοσύνης. Καλό όμω αυτό. Ήταν πολύ πλήρες και περιεκτικό ω παρέμβαση. Ναι, το λέω ως έπαινο. Ναι.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 Ευχαριστώ λοιπόν πολύ Κλοντ. Ευχαριστώ πρώτα για τις παρεμβάσεις από την Λετωνική Προεδρία πρώτα. Γνωρίζετε ότι δεν ήταν τόσο απλό κατά τη διάρκεια αυτού του εξαμήνου να μπορέσουν να προχωρήσουν πράγματα τα οποία επί μεγάλο χρονικό διάστημα είχαν παγώσει και δεν μπορούμε να αναμείνουμε ότι σε όλα θα υπάρχει πλήρης ικανοποίηση. Υπάρχουν και πολλές επικρίσεις ε, από την Ευρωβουλή ιδιαίτερα όσον αφορά την δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Τώρα, θεματολόγια, μερίσια διάταξη για τη μετανάστευση. Δεν μπορώ εγώ να εκφράσω την ικανοποίησή μου για μια τέτοια επιτυχία. Δεν είναι επιτυχία. Πόρο απέχει μια και μια ολόκληρη σειρά κρατών μελών και το δικό σας κράτος μέλος, η Λετωνία, είχαν πει ότι με την κατανομή των μεταναστών έχουν βλέπει προβλήματα και δεν υποστηρίζουν προτάσεις και τώρα αναφέρεται λέει ότι δεν θα είναι δεσμευτική μια τέτοια κατανομή και ακούσαμε ότι όλα αυτά λέει θα είναι μη δεσμευτικού χαρακτήρα. Ε τότε τι θα απογίνει στο τέλος τέλος με την Μέσια διάταξη για τη μετανάστευση. Έχουμε πολλές επικρίσεις. Αλλά αυτή τη στιγμή πώς έχει η κατάσταση σε σχέση με τα θέματα αυτά φοβούμε ότι δεν θα ληφθούν μεγάλες εμβέλειες αποφάσεις έχουμε επικρίσεις ε, έντονες και αυτές είναι εγκάρσιες ε, μέσω όλων των κοινοβουλευτικών ομάδων για αυτά τα θέματα ότι τα σκάφη των ε, λαθρεμπόρων, των ανθρωπεμπόρων θα καταστρέφονται και θα καταποντίζονται. Δεν υπάρχει όμως εντολή του, των Ηνωμένων Εθνών για μια τέτοια πρόταση και είναι κάτι το οποίο παραμένει μετέωρο σε σχεδιασμό και έτσι έχει διαδοθεί κάτι το οποίο δεν αξίζει τον λόγο να συζητείτε και ακολουθεί και μια λανθασμένη πορεία. Θα ήθελα να ακούσω το, την άποψή σας για το πώς έχει η στο Συμβούλιο από πλευρά των κρατών μελών για αυτό το θέμα και θα ήθελα να μου πείτε πώς εσείς στην ίδια σας τη χώρα, τη Λετωνία, αντιμετωπίζετε αυτά τα θέματα της μετανάστευσης που, δεν, τα υποστηρίζετε στις προτάσεις που έχουν διατυπωθεί κιόλα. Και τώρα σε σχέση με τις συμφωνίες και τις συνθήκες, ξέρετε ότι υπάρχει έντονη κριτική από την Ευρωβουλή. Για παράδειγμα, για το θέμα του Χαρτούμ και την δίκη του, ε, ε, του Ομάρ ε, Μπασίρ και όπως ξέρετε οι συνθήκες με άλλες χώρες όπως ε, για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης τούτων δεδομένων είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και υπάρχει και κάποια συζήτηση από πλευράς της ε, Ιταλικής κυβέρνησης που ξεκίνησε με προτάσεις της ε, και στο Συμβούλιο να τροποποιηθεί η Συμφωνία του Δουβλίνου, να αλλάξει το πλαίσιο της Συμφωνίας Δουβλίνου, γιατί και η Ιταλία, όπως επίσης εξάλλου και η Ελλάδα, έχουν σοβαρότατες επιφυλάξεις για τη διατήρηση και συνέχιση του συστήματος της Συμφωνίας του Δουβλίνου, που δεν μπορεί να γίνει με αυτόν τον τρόπο. Έχετε έστω και μία μόνο φορά συζητήσει τα θέματα των νόμιμων διάβλων και οδών μετανάστευσης προς την Ευρώπη για αυτούς τους μετανάστες. Έγινε ποτέ συζήτηση για μια ανθρωπιστική θεώρηση διαβατηρίου. Έγινε συζήτηση για παράδειγμα για τις νόμιμες οδούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση Μετανάστευσης. Για σας δεν διαδραματίζει αυτό κάποιο ρόλο. Παραμένετε μόνο στην καταπώντηση, στην βήθηση πλοίων και μόνο στη διατήρηση της Συμφωνίας του Δουβλίνου τι γίνεται σχετικά με εσά. Μια συγκεκριμένη ερώτηση θέλω να διατυπώσω και θέλω οπωσδήποτε να την απαντήσετε. Δεν ξέρω τι θα κάνετε με τι άλλε απαντήσει, αλλά αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να απαντήσετε. Η Ελλάδα θέλει, η νέα κυβέρνηση τη Ελλάδα θέλει να αλλάξει την πολιτική για τη μετανάστευση και το σύμφων, τις συμφωνίες πλαίσια. Και τώρα στην Ελλάδα υπάρχουν μόνο, υπάρχει στην Ελλάδα μια φυλακή εντό εισαγωγικών φυλακές στις οποίες ε, εγκαθίστανται αυτοί οι μετανάστες. Αυτές οι φυλακές, αυτά τα κρατητήρια θα κλείσουν. Όμως οικοδομήθηκαν με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γνωρίζουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα μπορούσε να ηγερθεί το αίτημα. Αυτά τα κονδύλια για την, για την έγερση, το χτίσιμο αυτών των φυλακών και κρατητηρίων να επιστραφούν λέει από την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι γίνεται με όλη αυτή τη συζήτηση. Όταν λέγεται ότι τα κράτη-μέλη υποστηρίζουν λέει στα θέματα μετανάστευσης, στα αιτήματα αυτά. Ερώτημα, αυτό αφορά όλα τα κράτη-μέλη ή μόνο κάποια λίγα και ανήκει και η Ελλάδα σε αυτά τα κράτη. Επίσης, Χαίρομαι βέβαια το ότι κάτι, σε κάτι καταλήξαμε. Έγινε λόγος για την 15η Ιουνίου. Πέρασε η 15η Ιουνίου και παραμένει λέει αυτή η τοποθέτηση επιθεμάτων αρχής και με ικανοποιεί αυτό. Όμως η μεγάλη μου ανησυχία είναι η οδηγία. Ξέρετε ότι θέλουμε να έχουμε μια δέσμη μέτρων που θα ισχύει. Θέλω να μου πείτε τι γίνεται με την οδηγία αυτή. Μπορείτε να, μου πείτε, να μας πείτε δυο λόγια κάτι παραπάνω δηλαδή για αυτήν. Ένα τελευταίο σημείο του οποίου δεν αναφέρθηκε τίποτα και υπάρχουν πολλά θέματα είναι το θέμα της NSA, της Αμερικανικής Υπηρεσίας Εθνικής εθνικής ασφάλειας National Security Agency και την παρακολούθηση πολιτών και μάλιστα με τη βοήθεια μυστικών υπηρεσιών άλλων κρατών μελών όπως δηλαδή εδώ της Γερμανίας. Υπάρχει μια έκθεση επ' αυτού ήδη από την τελευταία κοινοβουλευτική θητεία για τα θέματα παρακολούθησης. Σας ερωτώ γιατί δεν υπάρχουν κάποια συμπεράσματα από πλευρά του Συμβουλίου για αυτό το θέμα και σε σχέση με αυτό το πλέγμα, δηλαδή κατασκοπίας και παρακολούθησης από την NSA, όπως είχε κατά το παρελθόν τεθεί. Τώρα θα έχουμε και ένα ψήφισμα για αυτή την υπόθεση, που θα έχει όμως ως ε, περιεχόμενο επιτέλους να δράσουμε, γιατί δεν έγινε τίποτα μέχρι τώρα. Διαρωτώ με, πώς έχει συζήτηση στο Συμβούλιο για αυτά. Ευχαριστώ, Κορνίλια. Η Τζουδίθ Σαρτζεντίνη, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Παρακολούθησα τη συνέντευξη τύπου χθες το απόγευμα του Υπουργού Εσωτερικών Υποθέσεων. Είπατε χθες ότι συνομιλήσατε με τους συναδέλφους σας για πέντε ώρες για τη μετανάστευση. Σήμερα το πρωί είπατε ότι μιλήσατε για έξι ώρες. Ε, εν πάση περιπτώσει η έκβαση είναι φτωχή θα έλεγα τη συζήτηση. Είμαι λίγο απογοητευμένη ή μάλλον να το ξαναπώ, είμαι πάρα πολύ απογοητευμένη γιατί στο Κοινοβούλιο έχουμε συζητήσει για τη μετανάστευση και το άσυλο ξανά και ξανά και ο Επίτροπος Αβραμόπουλος μας λέει συνεχώς να είμαστε υπομονετικοί. Θέλει να προσπαθήσει, θέλει να προχωρήσει, αλλά πρέπει να λάβει υπόψη του ότι το κράτη-μέλη έχουν δυσκολίες να προσαρμόσουν την προσέγγιση τους και το καθεξής. Τα λέω αυτά με δικά μου λόγια, γιατί δεν ξέρω πραγματικά εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να κάνει τολμηρά βήματα. Έτσι ερμηνεύω όμως τα λόγια του Επιτρόπου Αβραμόπουλου. Είναι περίεργο να βλέπει κανείς και πρέπει να το πω ξεκάθαρα ότι η Ευρώπη είναι μια κοινωνία που γυράσκει. Έχουμε συγκρούσεις γύρω από τα σύνορά μας. Μπαίνει κόσμο στην Ευρώπη που είναι πολιτικοί πρόσφυγες και χρειάζονται ένα ασφαλές μέρος και μπαίνουν άνθρωποι στην Ευρώπη γιατί ζητούν άσυλο και γιατί ζητούν άσυλο γιατί δεν έχουν άλλη δυνατότητα, δεν μπορούν να ζητήσουν κάτι άλλο. Και εσείς δεν είστε έτοιμοι να καταλήξετε σε συμφωνία για την ανακατανομή των 40.000 ε, ανθρώπων που είναι στην Ευρώπη ήδη και την υποδοχή 20.000 ανθρώπων που είναι στα στρατόπεδα του ΟΗΕ στην άλλη πλευρά των ε, συνόρων. Έχουμε και πρέπει να έχουμε εργασιακή μετανάστευση σε μια κοινωνία που όλο και περισσότερο γυράσκει. γυράσκει. Και αν δεν είστε έτοιμοι να το κάνετε αυτό και να υποβάλλετε προτάσεις για να καταπολεμήσετε την παράτυπη μετανάστευση, αν το κάνετε αυτό χωρίς να είστε έτοιμοι να υποβάλλετε προτάσεις για την υποδοχή των ανθρώπων που χρειαζόμαστε, ε, τότε όλο και περισσότεροι θα μπαίνουν παράτυπα, θα είναι σε άσχημη κατάσταση, θα δουλεύουν σε φρικτές συνθήκες, θα επέφτουν οι τιμές της αγοράς, κάτι το οποίο είναι, θα είναι κακό για αυτούς αλλά και για τις δικές μας κοινωνίες. Πρέπει να κάνουμε αποτίμηση των αναγκών μας, να ξέρουμε τι χρειαζόμαστε και να δράσουμε και τα 28 κράτη-μέλη να αναλάβουν την ευθύνη τους. Συνοπτικά κύριε, το δικό σας εξάμεινο ήταν αργό. Ήσασταν αργοί και δεν καταλάβατε πόσο μεγάλη ήταν η κρίση που αντιμετωπίζουμε. Τελική ερώτηση. Μιλήσατε για αυτή τη διαδικασία Α, την διαδικασία Amberlight. Θέλω να μας πείτε περισσότερα. Ευχαριστώ. Ε, ο Πρόεδρος. Θα ήθελα και εγώ να πω κάτι. Ξέρετε, να σας πω μια εμπειρία που έχω, την εμπειρία που έχω από το 99. Μερικές φορές όταν σχολιάζουμε μια προεδρία μιλούμε για το κράτος μέλος και την έλλειψη διαφάνειας ή την κολυσιεργία. Όμως η προεδρία προσπαθεί να κάνει το διαιτητή μεταξύ των διαφορών συμφερόντων. συμφερόντων. Ε, θέτουμε το ερώτημα, τι συνέβη την Τρίτη, ποιος είπε τι δεν υπάρχει αρκετή διαφάνεια. Ό,τι πολιτική άποψη και να έχετε, δεν είπαμε ότι είναι κακή. Είπαμε ότι θέλουμε να ξέρουμε ποιο λέει τι. Δηλαδή, έγινε εγκρυπτό, αν θέλετε. Πρέπει σε μια συνέντευξη τύπου ένα υπουργό να μπορεί να το πει αυτό το πράγμα. Εμένα μου θέτουν αυτό το ερώτημα. Είναι δύσκολο γιατί εσείς είστε έχετε την Προεδρία και πρέπει να επιδείξετε διπλωματικές δεξιότητες, διοικητικές δεξιότητες. Ε, δεν προχωρούμε αρκετά γρήγορα, αναφέρεστε στο Amber Light στη διαδικασία αυτή. Είναι δύσκολη η θέση, θα σας το καταλαβαίνω. Είναι μια κατάσταση απογοητευτική. Εγώ υποτίθεται ότι μπορώ να πάω στα άτυπα συμβούλια, αλλά δεν μπορώ να πάω στα επίσημα συμβούλια υπουργών. Είναι μια κατάσταση απογοητευτική για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία μα ματαιώνει εμά εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συντούμε περισσότερη διαφάνεια, δεν ασκούμε κριτική για τι εκάστοτε πολιτικέ απόψει. Το επαναλαμβάνω ότι είναι ενοχλητικό, είναι απογοητευτικό. Δεν ισχύει βέβαια για όλε τι ε, προεδρίες. Η Κατερίνα και επανερχόμαστε στου υπουργού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε για το, το χρόνο ομιλίας που μου δίνετε. Να τον αξιοποιήσω ευχαριστώντας και εγώ την Προεδρία για τη δουλειά που έκανε και τους τριμερείς ε, διαλόγους για την οδηγία περί ενηλίκων. Πραγματικά έχει γίνει δουλειά με πολύ σοβαρή ε, εξέταση της ίδιας της οδηγίας και με σημαντικά σοβαρά αποτελέσματα για ένα θέμα όπου, όπως και τα άλλα που ως τώρα αναφέρθηκαν, υπάρχουν πολλοί ενδιασμοί, πολλά επικριτικά σχόλια και δεν είναι εύκολα, εύκολο να καταλήξουμε σε συμβιβασμό. Ευχαριστώ λοιπόν και πάλι την Προεδρία για τη συμβολή της. Παραμένοντας στο θέμα των ανηλίκων, είναι σημαντικό να τονίσω και το εξή. Τους μία συνόδευτους αλλοδαπούς ανηλίκους και ιδίως τους ε, ανηλίκους μετανάστες. Εδώ νομίζω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα. Οπωσδήποτε υπάρχει ανάγκη να γίνονται καλύτεροι έλεγχοι. Με περισσότερη συλλογή δεδομένων για αυτούς τους ανηλίκους. Για να αποφύγουμε, όπως συχνά συμβαίνει, να χάνονται αφού γίνει είσοδο στην επικρατεία μας και να είναι θύματα του οργανωμένου κλίματος, κάποιας μορφής ε, εκμετάλλευσης, όπως σεξουαλικής, ή από κυκλώματα ναρκωτικών και ούτω καθεξής. Για να μην πω ότι μπορούν να τους καταπιούν τα, τα πλοκάμια και τα δίκτυα τρομοκρατίας. Στο πολύ σύντομο λοιπόν χρόνο που έχει η Προεδρία σας, δεν θέλετε να δώσετε μια όθηση στο θέμα αυτό, μια επιπλέον όθηση, Λόγου χάρη προσαρμόζοντας και διευρύνοντας το σύστημα ΣΥΣ το σύστημα αυτό ελέγχου για να έχουμε πολύ συγκεκριμένα δεδομένα ώστε να μην χάνονται αυτοί οι ανήλικοι από τον έλεγχό μας. Και τα ζητήματα που επεσήμεναν οι συνάδελφοι ήταν όλα πάρα πολύ σημαντικά, αλλά δεν θέλω να επεκταθώ για να υπάρξει χρόνος για τις απαντήσεις. Παρ' όλα αυτά, έγινε λόγος και για ένα πολύ σημαντικό για μας ζήτημα, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ποιες είναι οι περαιτέρω προοπτικές για το θέμα αυτό. Ε, στο σημείο όπου φτάσαμε με την Λετωνική Προεδρία και ένα άλλο θέμα, ένα σημαντικότατο θέμα των εφιών συνόρων. Το συζητήσαμε το θέμα αυτό. Έχει γίνει ανάλυση κόστους ωφελίας. Το κόστος είναι υψηλό και θα πρέπει να έχουμε όλα τα στοιχεία που θα μας επιτρέψουν να αποτιμήσουμε σωστά την αποτελεσματικότητα του συστήματος αυτού. Ακόμη ένα θέμα, πάω λίγο πίσω, ξεπερνώντας κάποια άλλα επίσης σημαντικά ζητήματα, μετανάστευση. Σημαντικές παρατηρήσεις και από τους συναδέλφους και δεν μπορώ να παραγνωρίσω. Εγώ έρχομαι από τη Σικελία. Η επικράτειά μας πλήττεται με τρόπο δραματικό και συστηματικό από το φαινόμενο της μετανάστευσης. Τόσοι απελπισμένοι που διασχίζουν τη Μεσόγειο και ξεβράζονται ή τέλος πάντων διασώζονται στις θάλασσες της Σικελίας. Είδαμε να πνίγονται πολλές φορές μπροστά στα μάτια μας σχεδόν, στις ακτές μας. Είναι πολύ δραματική η διάσταση αυτού του θέματος και διαρωτώ Υπόθηκαν τόσα πολλά, όμως υπάρχει και κάτι άλλο που δεν μπορώ παρά να υπογραμμίσω. Υπάρχει μια αντίφαση μεταξύ της δράσης των τρομοκρατικών ομάδων που ε, στηρίζουν αυτές τις μετακινήσεις, την εμπορία των μεταναστών και αποσπούν τεράστια οικονομικά ωφέλη από αυτή την εμπορία. Τι μπορούμε να κάνουμε, χωρίς να παραγνωρίζουμε όλες τις άλλες πτυχές που τονίστηκαν. Πιστεύω το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρόεδρος, ευχαριστούμε Κατερίνα. Θα κλείσω τον κατάλογο των αγορητών γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί που πήραν τον λόγο. Κύριε Τσάκη, παρακαλώ. σε ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, δύο λόγια μόνο θα ήθελα να πω. Κατανοώ και η κριτική και οι επικρίσεις από τους ευρωβουλευτές οφείλονται στο ότι υπήρξαν ε, προβλήματα στην αντιμετώπιση των θεμάτων μετανάστευσης. Δεν συμφωνώ όμως όλα αυτά ότι πρέπει να διοχετευτούν κατά της Λετωνίας ως ε, χώρας που άσκησε την Προεδρία. Δεν αντέδρασε με ταχύς ρυθμούς η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ούτως έχουν τα πράγματα σε σχέση με την, ε, με την δομή των θεσμικών οργάνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έπρεπε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών να εμπλακούν περισσότερο περισσότερο. Δεν είναι δυνατόν τα θέματα μετανάστευσης να επιληθούν αποκλειστικά στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ανατολική Αφρική και στην ε, Μικρά Ασία πρέπει να αναλυθούν πρωτοβουλίες. Εξαιρετική ήταν η συνεργασία αυτό το εξάμεινο και με τους δύο από εσά υπουργού. Ε, και σε σχέση με τον τριμερή διάλογο και το ανέφερε και η Καταδίνα οι επιδόσεις της Προεδρίας σας ήταν ιδιαίτερα αξιόλογες και και η ανακυκλούμενη εξάμεινη προεδρία είναι κάτι το οποίο μπορεί να εξηγήσει πολλές φορές ε, σε τι οφείλονται κάποια προβλήματα. Και ευχαριστώ για τις ε, ερωτήσεις και τις απαντήσεις ε, που δόθηκαν. Ξεκινάμε τώρα με την παρέμβαση του Υπουργού. Ξεκινάμε τώρα με αυτή τη σειρά. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις που διατυπώθηκαν. Οι περισσότερες από τις ερωτήσεις συνδεόντουσαν με προβλήματα μετανάστευσης τα οποία αντιμετωπίζουμε και πρέπει να επιληθούν. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ένα γενικότερο πλαίσιο, γιατί κάθε ερώτηση και κάθε ευρωβουλευτής ανέφερε το θέμα της μετανάστευσης σε κάθε παρέμβαση αναφύεται το θέμα λοιπόν της μετανάστευσης. Δεν κοίταξα το ρολόι μου ακριβώς και δεν, ε, δεν μπορώ να σας ε, πω ε, ποια ήταν ακριβώς η διάρκεια όλων αυτών. Όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι προτάσεις της οι προτάσεις αυτές γνωστοποιήθηκαν κατά την 13η Μαΐου. Είχαμε την πρώτη συζήτηση σε επίπεδο Υπουργών στο Συμβούλιο με συμμετοχή όλων των κρατών. Οι εταίροι μας ε, συμμετείχαν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και για τον Ευρωπαϊκό ε, Οικονομικό Χώρο μπορούν να διατυπωθούν ε, οι λύσεις που προτείνονται σε τρεις άξονες ε, βραχυπρόθεσμους άξονες, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους έγινε μια παρέμβαση σε σχέση με την αντιμετώπιση των σκαφών και των λαθρεμπόρων η καταπολέμηση των ανθρωποεμπόρων και λαθρεμπόρων δεν θα σημαίνει ότι θα βυθίζονται τα σκάφη αυτά με τους ε, πρόσφυγες, με τους μετανάστες ε, μέσα στα σκάφη αυτά. Θα θέλαμε όμως να καταστραφούν, να καταστρέφονται τα σκάφη αυτά προτού επιβιβαστούν σε αυτά οι μετανάστες, οι πρόσφυγες. Είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα. Δεν μπορούμε όμως να αγνοήσουμε αυτό τον συντελεστή, αυτή την παράμετρο, επειδή είναι μια ε, κατέγινε πλέον, κατέληξε στο να είναι μια πάρα πολύ κερδοφόρος επιχείρηση αυτή η μεταφορά των ατόμων αυτών. Εκατομμύρια αποκομίζουν οι εμπλεκόμενοι λαθρέμποροι και πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Συνεργασία με τρίτα κράτη. Είμαστε ότι χωρίς συνεργασία με τα τρίτα κράτη θα αυξηθούν αυτές οι μεταναστευτικές ροές. Και τώρα να γνωρίζουμε το πόσα άτομα είναι διατεθειμένα να ξεκινήσουν ένα τέτοιο επικίνδυνο ταξίδι που γνωρίζουμε ότι πρέπει να γίνει λόγος για εκατομμύρια ε, φιλόδοξων τέτοιων μεταναστών, επίδοξων μεταναστών και πρέπει να αναλυθούν όλα εκείνα τα μέτρα για να είμαστε σε θέση να αποκατασταθεί, να εξευρεθεί μια ισορροπία μεταξύ των πραγμάτων και να εξομαλυνθεί η κατάσταση και στις ίδιες τις χώρες από τις οποίες υποχρεώνονται αυτοί οι άνθρωποι να ε, τις εγκαταλείψουν και να διαφύγουν από εκεί. Τώρα, για το, τα μέτρα τα οποία προτάθηκαν και την υποστήριξη σε αυτά, δεν μπορώ τώρα ακριβώς να σας αναφέρω ποια ήταν ακριβώς η πρόταση και η παρέμβαση της κάθε χώρας. Μπορείτε να στραφείτε βέβαια στις κυβερνήσεις σας και να τις ρωτήσετε ποιες ήταν οι παρεμβάσεις της και οι συνεισφορές από πλευράς της. Όμως μπορώ να αναφέρω σε σχέση με το αν η προσέγγιση αυτή θα πρέπει να είναι υποχρεωτική, δεσμευτικού χαρακτήρα ή μη δεσμευτική, <clears throat> εθελούσιου χαρακτήρα και άλλες εναλλακτικές λύσεις συζητήθηκαν για την κατανομή, για παράδειγμα για μια κλίδα κατανομής ε, ε, προσφύγων και θα ήθελα να αναφέρω ότι αυτή η συζήτηση διεξήχθη χωρίς καμιά καθυστέρηση, άμεσα και βρισκόμαστε σε μια κατάσταση και κινούμεθα προς το η αρχή της αλληλεγγύης να μπορεί να είναι σεβαστή και να εφαρμόζεται. Εμένει και επιμένει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επ' αυτού και πιστεύω, ευελπιστώ ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμό κατά τους επόμενους μήνες. Ιδιαίτερα για να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε τα, τις χώρες ε, της πρώτης γραμμής, ε, τις χώρες που βρίσκονται στο μέτωπο αντιμετωπίζοντας τις, τους μετανάστες αυτούς όπως την Ελλάδα και την Ιταλία. <clears throat> Θα ήθελα να πω ότι όπως ακούστηκε προηγούμενα και η Λετωνία αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις σας εμείς δεν καθυστερήσαμε ως λεπτονική προεδρία με κανένα τρόπο τα πράγματα. Συνοψίσαμε το πώς έχουν ε, τα πράγματα, πώς εξελίχθηκε η κατάσταση. Θα δώσουμε τη σκητάλη της προεδρίας στο Συμβούλιο πολύ σύντομα στο Λουξεμβούργο και το θέμα αυτό θα ε, επανέλθει στην ημερήσια διάταξη των θεμάτων υποσυζήτηση συντομότατα. Όσον αφορά το κέντρο κατά της τρομοκρατίας και την Europol την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία και <clears throat> θα στόχος του κέντρου θα είναι να συντονίζονται οι πληροφορίες και η χρήση των πληροφοριών αυτών με τον βέλτιστο τρόπο. Η διάχυση και η διαχείριση ε, λειτουργικά αυτών των πληροφοριών διότι γνωρίζουμε ότι σε αρκετές χώρες υπήρξε παράνομα, υπήρξαν παράνομα δίκτυα ε, όπλων και οπλισμού και οι πληροφορίες ε, της Ευρωπόλ μπορεί να είναι πολύ επικοδομητικές. Όσον αφορά το κέντρο για ε, τις έρευνες δεν ήταν δυνατόν να επιτευχθεί το μέγιστο αποτέλεσμα. Κάναμε όμως ό,τι ήταν εφικτό για να σημειωθεί πρόοδος στο πεδίο αυτό. Και όσον αφορά την ΣΥΠΟΛ και τις διατάξεις για την ΣΥΠΟΛ και την Europol, κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας για να σημειωθεί πρόοδος ε, στα θέματα. Τώρα, σε σχέση με την Συμφωνία Δουβλίνου και την τροποποίηση ή μεταρρύθμιση του συστήματος. Διεξήχθησαν συζητήσεις στο Συμβούλιο επ' αυτού και αναμένουμε αυτή τη στιγμή να υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρότασή της από πλευράς της και μπορώ να επιβεβαιώσω ότι συζητήσαμε όλα τα θέματα που αφορούν την μετανάστευση και την επανεισδοχή, θέμα το οποίο ιδιαίτερα συζητήθηκε κατά τη διάρκεια του γεύματος εργασίας που είχαμε υπήρξε και μια συζήτηση για το Amber Light και την διαθεσιμότητα των στοιχείων. Μπορώ να επαναλάβω σε σχέση με τα δεδομένα αυτά τα οποία προανέφερα. 28 κράτη-μέλη συμμετείχαν σε σχέση με πληροφορίες από 55 αερολιμένες, 55 αεροδρόμια και υπήρχαν ανησυχίες λύματα ότι κάποια άτομα τα οποία είχαν παραβιάσει την διάρκεια της ε, θεώρησης ε, διαμονής που είχαν ε, θα συλλαμβάνονται. Ωστόσο κανείς δεν συνελήφθη και εν συντομία αυτά είχα να σας πω και θα δώσω τον λόγο στον συνάδελφό μου. Yes, please go ahead. Παρακαλώ, Υπουργέ. Πολλοί είναι συνάδελφοι που με γραπτά μηνύματα με ειδοποιούν ότι ζητούν συγγνώμη που δεν μπορούσαν να έρθουν σήμερα, αλλά υπήρχαν δυσκολίες με τις ε, ταξιδιωτικέ τους ε, διευθετήσεις. Ε, ζητούν λοιπόν συγγνώμη. Θα υπήρχαν περισσότεροι παρόντες. Ξέρω ότι πολλοί έχουν συνεργαστεί μαζί σας στους τριμερές διαλόγους, με τους συνεργάτες σας είναι γι' αυτό και μόνο το λόγο χαμηλότερη προσέλευση σήμερα. Παρακαλώ κύριε Υπουργέ. Έχετε χρόνο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τους ε, βουλευτές ε, για τις ε, για τις παρατηρήσεις τους. Ε, για την πρόοδο στον κανονισμό κατά την οδηγία ε, και τα σχόλια ότι ήταν ανεπαρκής. Να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να δώσω κάποιες πρόσθετες πληροφορίες. Η κυρία Σίπελ ρώτησε εάν η οδηγία θα εγκριθεί τον Οκτώβριο. Στις 24 Ιουνίου έχουμε προγραμματίσει έναν τριμερή διάλογο εδώ και εντός αυτού του τριμερούς διαλόγου, το Λουξεμβούργο θα σας ενημερώσει για τις προτεραιότητές του. Μία από τις προτεραιότητές τους, εξ όσων γνωρίζω, είναι η έγκριση ακριβώς της οδηγίας, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου τους. Σε κάθε περίπτωση, είστε πρόσδεκτοι στην συνάντηση αυτή και θα ακούσουμε με ιδιαίτερη προσοχή τις προτεραιότητες του Λουξεμβούργου που έχουν ανακοινωθεί από τις 25 Μαΐου στο Λουξεμβούργο αλλά και κατά την άτυπη των Ηνωμένων Πολιτειών με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία ακόμη ερώτηση τέθηκε για το τι πρόοδος έχει επιτευχθεί και γιατί αργούμε. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε αν δεν υπάρξει μια γενική ε, προσέγγιση που να έχει εγκριθεί. Ρωτήθηκε και άλλοι το ρώτησαν Τι μπορεί να γίνει για αυτό το ζήτημα παράλληλα με άλλα. Ο κανανισμός αφορά τα ζητήματα των πολιτών και η οδηγία την ποινική διάσταση. Υπάρχουν 91 άρθρα σε 250 σελίδες για να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ 28 κρατών μελών για την διατύπωση δεν είναι κάτι απλό. Πόσες συναντήσεις φαντάζεστε ότι χρειαστήκαμε αυτούς τους μήνες για να συζητήσουμε άρθρο προς άρθρο και να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα. 45 συναντήσεις χρειάστηκαν. Και να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονες που έκαναν σχεδόν πραγματικότητα το αδύνατο. Πολύ αντιφατικές απόψεις, από τη μια εμπειρογνώμονες και από την άλλη ε, πολιτικοί ε, πρόσωποι που ήθελαν να ε, καταλήξουν σε πλειοψηφία. Ήταν αδύνατη αποστολή αυτό που επιτύχαμε. Αλλά τα καταφέραμε. Και είμαστε πολύ περήφανοι. Σε ό,τι αφορά την οδηγία και τον κανονισμό λοιπόν, έγιναν και άλλες ερωτήσεις για τα θέματα αυτά να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής σας που συνεργάστηκαν μαζί μας στους τριμερείς διαλόγους, ιδίως την κυρία Κινίτσι, για την ε, ιδιαίτερα επικοδομητική συνεργασία για τις ε, δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά. Τα δεδομένα αυτά νομίζω μας επιτρέπουν να υποθέσουμε ότι οι τριμερείς διάλογοι θα προχωρήσουν ε, θετικά. Πρόεδρος, ευχαριστούμε τους υπουργού, σας ευχαριστώ συνάδελφοι και πάλι καθώς είναι το τέλος της προεδρίας σας, εκ μέρους όλων των συναδέλφων και όσων είναι παρόντες και όσων είναι απόντες, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη σκληρή σας δουλειά. Εσάς και όλους σας τους συνεργάτες. Κάποιους από εσά τους γνωρίσαμε το τελευταίο εξάμεινο και πραγματικά ε, αισθανόμαστε ευγνωμοσύνη για όσα κάνατε, για τη διοργάνωση των συναντήσεων και το καθεξής και για το σεβασμό τον οποίο μας δείξατε. Ήταν ένα υπέροχο εξάμεινο. Και πιστεύω ότι θα παραμένουμε σε επαφή και μετά από αυτό το εξάμεινο. Thank you.